ευχαριστήσω εκ νέου τους συναδέλφους για τις προτάσεις τους. Κάποιες τροπολογίες που θεωρώ ότι δεν μπορούν να γίνουν δεκτές, ενδεχομένως μετά τη συνάντησή μας να επιτρέψουν να επέλθει κάποια συμφωνία με τους συντάκτες των τροπολογιών, γιατί πιστεύω ότι επί της ουσίας συμφωνούμε. Ίσως ο τρόπος έκφρασης να είναι κάπως λάθος με την ότι είτε παρά είναι ε, συγκεκριμένες είτε παρα, παρα είναι ρητές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σχόλια. Κύριο Ζαλέτσκι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το ΕΛΚ, Ευρωπαίοι Δημοκράτες, και εγώ προσωπικά μπορώ να σας πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος με τις αλλαγές της συγγήτριας για τα σχολικά εγχειρίδια στο γυμνάσιο και το λύκειο ούτως ώστε να μπορούμε να αναδείξουμε τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το λόγο γένεσής της με καλύτερο τρόπο μεταξύ των μαθητών, ούτως ώστε η κοινωνία ευρύτερα να καταλαβαίνει τι στόχο έχει η Ένωση. Η τροπολογία 13 ε, την έχει απορρίψει η συγγήτρια. Βασίζεται σε μια προσωπική εμπειρία μου όταν οργάνωνα διάφορες πρωτοβουλίες όχι σε σχολεία κατά ανάγκη. Ωστόσο ε, μερικές φορές αυτές οι πρωτοβουλίες ε, πραγματοποιούνται από μαθητές και βοηθούν να αυξηθεί η συνειδητοποίηση στην κοινωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλώ για τις τοπικές πρωτοβουλίες σε πόλεις και κομοπόλεις όπου οι μαθητές προσπαθούν να κινητοποιήσουν τον τοπικό πληθυσμό, την αστυνομία, το Δήμο, τις τοπικές αρχές, τη, τους ιερείς, τους τοπικούς επιχειρηματίες για να συμμετάσχουν σε τέτοια προγράμματα. Μέσω της, ε, των προγραμμάτων αυτών ο κόσμος μαθαίνει περισσότερα για την Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή εμπλέκεται προσωπικά. Έχω την άποψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αναλάβει κάπως το κόστος. Δεν είναι τζάπα όλα αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν δώσουμε κάποια κονδύλια στα έργα αυτά δεν θα είναι κακή ιδέα. Το να δώσουμε δηλαδή χρήματα σε κάποιες οργανώσεις που ξέρουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει νόημα. Ε, καλύτερα να δώσουμε κονδύλια κοινοτικά σε τέτοιες πρωτοβουλίες. Αυτά ήθελα να πω για τα σχολεία εν γέννη. Σε ό,τι αφορά ιδίω τις τοπικέ πρωτοβουλίες, ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε συνάδελφοι, θέλω να υποστηρίξω την τοπολογία 5, δική μου τοπολογία. που αφορά στο λεγόμενο δημοκρατικό κενό, όχι έλλειμμα, έτσι το λέμε εμείς στην ε, Συνταγματική Επιτροπή. Έλλειψη νομιμοποίησης της Ένωσης από τους πολίτες. Πρόκειται για μια τεράστια πρόκληση και ένα μεγάλο πρόβλημα. Προχωρούμε, πετυχαίνουμε πολλά, ωστόσο δεν πάει η επαφή με τον πολίτη. Η τροπολογία μου, έτσι είπε η συγκήτρια, θέλει να ε, μπει και χωρισμένα Δεχόμαστε ότι υπάρχει έλλειψη επαφής, αλλά θέλουν οι συγκίτρια από την άλλη πλευρά να ε, διαγράψει την διαπίστωση ότι πρόκειται για ένα μεγάλο πρόβλημα με τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και τα μέσα που δεν μας βοηθούν και που δύσκολο μπορούμε να παρακινήσουμε ώστε να έρθουν να βοηθήσουν την επαφή των ευρωπαϊκών οργάνων με τους πολίτες. Ενώ επιπλέον υπάρχει και το πρόβλημα της διαβούλευσης με τους πολίτες. Προτείνεται να υπάρξει ένας νέος οργανισμός. Αυτό το είχαμε συζητήσει στα πλαίσια της Επιτροπής ΑΦΚΟ συνταγματικών υποθέσεων, συζητήθηκε χτες, εκτιμήθηκε θετικά από την Επιτροπή και επί του θέματος αυτού θα γίνει μια συζήτηση τον άλλο μήνα στο Στρασβούργο. Παρακαλώ λοιπόν συνάδελφοι να υποστηρίξετε αυτό το κείμενο που θα βοηθήσει και την έκθεση Χέγγι γιατί Ένα βασικό πρόβλημα επαφής με τον πολίτη είναι αυτό του ρόλου και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των μέσων και δημιουργώντας άμεση επαφή μεταξύ πολίτη και θεσμικών οργάνων. Κάτι βασικό για να προχωρήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. <clears throat> Θα ήθελε να παρέμβει ίσως η Κομισιόν. Κύριε Γιώγνε, θέλετε να λάβετε τον λόγο. Η Κομισιόν. Όχι, δεν θέλουμε. Δεν έχουμε κάποιον να σχολιάσει. Δεν βλέπω κάποιο συνάδελφο ο οποίος να θέλει να μιλήσει σηκώνουν το χέρι του. Ζητώ λοιπόν από την εισηγήτρια να κλείσει τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Σαλέσκη. Εμείς προσπαθήσαμε να έχουμε κάποιες τροπολογίες συμβιβασμού. Για την τροπολογία 13 όμως νομίζω ότι συμφωνούμε καταρχήν επί της ουσίας αλλά Ίσως είναι καθαρά προσωπική η άποψή μου στο σημείο αυτό, αλλά πιστεύω ότι σε κάθε εκθέση που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ο στόχος μας είναι κάθε φορά να επανεφεύρουμε τον τροχό. Έχουμε πάρα πολλές ιδέες, προτάσεις, νέες ε, συστάσεις που ουσιαστικά μπερδεύουν πάρα πολύ τις εργασίες μας, περιπλέκουν και τη ζωή των πολιτών μας όταν θέλουμε να, όταν θέλουν να καταλάβουν τι ακριβώς κάνουμε. Γι' αυτό ο στόχος μου στο δικό μου έργο, όταν εγώ επεξεργάζομαι μία έκθεση, είναι το πώς θα μπορέσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα εργαλεία που ήδη έχουμε, τα ψηφίσματα που έχουμε και τις προτάσεις που έχουμε. Η Ετροπολογία 13 λοιπόν του κ. Σαλέσκη λέει ότι ζητάει από την Κομισιόν να δώσει μία μεγαλύτερη χρηματοδότηση για σχέδια τα οποία θα προωθήσουν τις ιδέες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμφωνώ με αυτή την έννοια, αλλά σίγουρα κανείς δεν ξέρει πολύ καλά ποιες είναι οι ιδέες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μου πείτε οι αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το καταλαβαίνω. Αυτό καταρχήν. Επιπλέον υπάρχουν ήδη προγράμματα τα οποία κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή και προωθούν τα θέματα αυτά. Υπάρχουν τα προγράμματα διαβίου εκπαίδευσης τα οποία είναι θαυμάσια και τα οποία είναι τα προγράμματα που ξεκινούν από το Κομμένιου στο, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, στο Λεωνάρντο, στη δευτεροβάθμια, Εράσμου κτλ. Είναι προγράμματα τα οποία λειτουργούν πάρα πολύ καλά. Αυτό το οποίο εγώ θα ήθελα να προτείνω λοιπόν είναι αντί να πούμε θα δημιουργήσουμε ένα νέο πρόγραμμα, όχι, να ζητήσουμε τα προγράμματα αυτά να έχουν καλύτερη χρηματοδότηση, να αυξηθεί η χρηματοδότησή τους. Με τον τρόπο αυτό θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα και αυτή θα πρέπει να είναι η θέση μας. Για το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας που λέει ότι τα προγράμματα αυτά θα πρέπει να προσανατολίζονται περισσότερο στους φοιτώντες στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση. Και έχει συνέπειες αυτό για τις τοπικές κοινότητες και αρχές δεν νομίζω ότι χρειάζεται να είμαστε τόσο επακριβεί στο θέμα αυτό και τόσο συγκεκριμένοι, γιατί όπω ξέρετε πολλά από αυτά τα θέματα τη εκπαίδευση είναι στην πραγματικότητα αρμοδιότητα των κρατών μελών και εμεί δεν μπορούμε να επιβάλλουμε, μπορούμε να προτείνουμε, να συνιστήσουμε, αλλά λειτουργεί καλύτερα αν δώσουμε γενικέ κατευθύνσει και όχι επιταγέ. Κατά τα άλλα μπορούμε να προσπαθήσουμε να συζητήσουμε να βρούμε μια λύση η οποία θα είναι ε, του ίδιου αποτελέσματος αλλά χωρίς να περιπλέξει περισσότερο το κείμενο της έκθεσης. αυτά που λέει ο κ. Μπιολογιεύσκη στην τροπολογία 5. Εδώ η αλήθεια είναι ότι το πρώτο τμήμα της τροπολογίας όπου εκφράζει την ανησυχία του για το χάσμα που υπάρχει μεταξύ των πολιτών της Ευρώπης και των θεσμών της Ευρώπης, αυτό είναι απόλυτα αποδεκτό από μένα. Γιατί αυτό δεν είναι μονάχα κάτι που λέμε εμείς είναι κάτι το οποίο το καταδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις, τα ευρωβαρόμετρα, οι έρευνες της Κομισιόν. Επομένως, από αυτή την άποψη συμφωνούμε. Αλλά μετά από αυτό το πρώτο τμήμα, λέει ο κ. ότι αυτό το χάσμα αντανακλάται από την έλλειψη ενδιαφέροντος που δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης και τα εθνικά κόμματα. Αυτό εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αιτιακή σχέση εδώ πέρα. Ίσως σε ορισμένε χώρες αυτό να ισχύει. Ίσως τα εθνικά κόμματα να ενδιαφέρονται περισσότερο και άλλα λιγότερο. Αλλά ότι όλα τα μέσα ενημέρωσης έχουν τέτοιο πρόβλημα, ούτε αυτό θα τολμούσα ποτέ να το πω. Θα χρειαζόμασταν περισσότερη βοήθεια από τα μέσα ενημέρωσης, ναι. Αλλά νομίζω ότι το να κάνουμε μια τέτοια συνολική διατύπωση δεν ευσταθεί. Τρίτο τμήμα της, της τροπολογίας, ο κ. Μπιαλοβιέσχη, ίσα τη δυνατότητα να υπάρχουν μηχανισμοί γενικευμένης διαβούλευσης με τους πολίτες, εγώ το βλέπω να είναι άκρος πεπλεγμένο αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή, αν πάνε όλα καλά, βρισκόμαστε πρώτων θυρών της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας στο τέλος του έτους ή στην αρχή του 2010. Ήδη η συνθήκη της Λισαβόνας προβλέπει τις ε, λαϊκές πρωτοβουλίες, προβλέπει μια σειρά από μέτρα τα οποία θα βοηθήσουν να υπάρχει μια πιο κοντινή σχέση με τους πολίτες. Επομένως, θα έλεγα ας θέσουμε σε εφαρμογή τη συνθήκη της Λισαβόνας το ταχύτερο δυνατό και ας δούμε μετά τι θα πρέπει να κάνουμε και μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις που ήθελα να κάνω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Η ψηφοφορία θα γίνει σήμερα το απόγευμα. Σας ευχαριστώ πολύ και περνάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, το υπαριθμό 12, απαλλαγή για το 2007, ε, τμήμα 3 του προϋπολογισμού και συντάκτης της γνωμοδότησης ο κύριος Ιστβαν Σαντιβάνη. Έχουμε μόνο δύο τροπολογίες. Όπως θα θυμάστε έγιναν κάποιες συζητήσεις για το θέμα αυτό, για τον έλεγχο του προϋπολογισμού ως προς τις δαπάνες για το Αφγανιστάν και το Ιράκ είτε απευθείας είτε μέσω οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών τα οποία αναφέρει και ο συντάκτης ε, στη γνωμοδότησή του. Να το δώσω λοιπόν το λόγο για μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Κύριε Σεντιβάνη, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα κάνω μια πολύ σύντομη περιγραφή της γνωμοδότησής μου. Έχουμε τέσσερα βασικά σημεία. Το πρώτο είναι ότι θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να βελτιώσει τη διαδικασία παρακολούθησης και παλήθευσης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο τομέας αυτός, κυρίως στο επίπεδο των οργανισμών που εφαρμόζουν και επίσης θέλουμε να μειώσουμε και το γραφειοκρατικό άχθος. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο περιμένω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το δεύτερο είναι πιο ευαίσθητο θέμα και εδώ έχουμε και τις δύο τροπολογίες που στοχεύουν σε αυτά τα δύο σημεία. Ζητάμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τις προσπάθειές της για να δώσει όλες τις πληροφορίες που έχουν δοθεί στο ελεγκτικό συνέδριο ε, που έχουν ζητηθεί συγγνώμη, από το ελεκτικό συνέδριο από τα Ηνωμένα Έθνη εγκαίρως. Ξέρετε ότι αυτό το θέμα διονύζεται συνεχώς, έχει γίνει μια κάποια πρόοδος και αναγνωρίζω και τη συμφωνία ΦΑΦΑ και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλή. Συμφωνία Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Ηνωμένων Εθνών. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να δούμε και τι γίνεται σε θέματα πρακτικής και εφαρμογή. Δηλαδή, να υπάρχουν αποστολές ε, οι οποίες θα επαληθεύουν ότι όντως ε, τίθενται σε πρακτική εφαρμογή και να βλέπουμε τι γίνεται. Θα πρέπει να υπάρχει διαφάνεια στην όλη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη και του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, διότι θεωρούμε ότι αυτή η τομή είναι σχετικά προβληματική. Τρίτον, καλούμε τις εθνικές αρχές να συμμορφωθούν με τους ε, κανονισμούς. Υπάρχουν ε, πολύ σοβαρά προβλήματα σε κάποιες χώρες με τους εφαρμοστικούς κανονισμούς, κυρίως ε, στη Βουλγαρία και στην Τουρκία και ελπίζουμε οι εθνικές αρχές να συμμορφωθούν προς αυτές τις απαιτήσεις. Και το επόμενο σημείο είναι ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περιμένει να ενημερώνεται τακτικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για, την, ε, ε για τις για την υποστήριξη της γεωργίας ε, μετά από την ε, σύραξη και θέλουμε να λαμβάνουμε τις πληροφορίες αυτές εγκαίρως και να είναι και αρκετά διεξοδικές ως προς το τι διαδικασίες ακολουθούνται. Τώρα, για τις δύο τροπολογίες. Η πρώτη τροπολογία αναγνωρίζει την πρόοδο που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι τούδε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό, το αναγνωρίζω, αλλά μπορώ να τη δεχτώ υπό την προϋπόθεση η τελευταία φράση της πρώτης παραγράφου να μην διαγραφεί. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τμήμα της γνωμοδότησης και δεν θα πρέπει να διαγραφεί. Δηλαδή, το without this leading to unnecessary administrative burdens for the end beneficiaries. Είναι πολύ σημαντική αυτή η φράση, θα ήθελα να παραμείνει. Κατά τα άλλα, μπορώ να δεκτώ ε, την ε, τροπολογία των Γκραφ ε, Λάμστρον κλπ. Τώρα, στη δεύτερη τροπολογία είμαι αντίθετος. Πιστεύω ότι αν δεχτούμε τη δεύτερη τροπολογία, να χρησιμοποιήσουμε τέτοια διατύπωση εξασθενίζει το τεράστιο πολιτικό μήνυμα του σχεδίου γνωμοδότησης, της γνωμοδότησής μου το βασικό μήνυμα και είμαι βέβαιος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρειάζεται να της αποστείλουμε ένα τέτοιο μήνυμα, όχι μόνο το Κοινοβούλιο, άλλωστε το Κοινοβούλιο είναι ο θεματοφύλακας των χρημάτων των φορολογωμένων. Επομένως θα πρέπει να διευκρινίσουμε, να είμαστε σαφείς ως προς το ότι υπάρχουν προβλήματα και πρέπει να γίνουν βελτιώσεις. Αν δεχτούμε αυτή τη δεύτερη τροπολογία, τότε εξασθενίζουμε και μάλιστα καταστρέφουμε και το ίδιο το μήνυμα που θέλουμε να αποστείλουμε αυτή τη γνωμοδότηση. Γι' αυτό λοιπόν είμαι κατά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σαντιβένη. Ο κύριος Γκάλερ. Ναι, ναι, ναι, uh, Συμφωνεί ο κύριος Γκάλερ, δεν χρειάζεται να μιλήσει, λέει. Άλλος κάποιος ο οποίος θα ήθελε να λάβει το λόγο η Κομισιόν ίσως. Ευχαριστώ Πρόεδρε, καλημέρα. Ευπρόσδεκτη έκθεση. Πράγματι, ανησυχούμε τα μάλα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε τα χρήματα του φορολογούμενου να χρησιμοποιούνται σωστά. Και αυτό σε όλα τα πλαίσια στα οποία κινούμαστε. Ο δημοσιονομικός κανονισμός δημιούργησε το σύστημα κοινής διαχείρισης. Βοηθάει. Νομίζουμε ότι η συμφωνία μας με τον ΟΗΕ είναι καλή. Βέβαια είναι πολύ μεγάλοι οργανισμοί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ΟΗΕ, άρα είναι αναπόφευκτο να υπάρχουν κάποια προβλήματα στην επαλήθευση και στον έλεγχο λόγω παρεξηγήσεων και κυρίως παρεξηγήσεων αφορά τον τρόπο λειτουργίας των λεκτικών μηχανισμών. Πιστεύουμε όμως ότι μπορούμε να εργαστούμε καλά με τον ΟΗΕ. Έγινε μια αξιολόγηση πρόσφατα, ήταν θετικότατη όσον αφορά την προστιθέμενη αξία που μπορούμε να κερδίσουμε διοχετεύοντας πόρους μέσω του ΟΗΕ κυρίως ε, σε περιστάσεις που εμείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα είμαστε θέση να χορηγήσουμε βοήθεια σε περιστάσεις μετά από καταστροφές, μετά από συγκρούσεις. Αυτή η συνεργασία με τον ΟΗΕ είναι σημαντικότατη για μας. Εξίσου σημαντικό είναι να έχουμε την πλήρη διαβεβαίωση ότι θα έχουμε πρόσβαση στα αναγκαία για την επαλήθευση. Συνήθως οι έλεγχοι διεξάγονται ομαλά. Δεν έχουμε γενικά πρόβλημα. Γίνεται αυξανόμενος έλεγχος των χρημάτων που διοχετεύονται μέσω του ΟΗΕ. Και συνήθως οι έλεγχοι πηγαίνουν καλά. Θέλουμε όλοι να πηγαίνουν καλά όμως οι έλεγχοι. Γι' αυτό συνεργαστόμαστε με τον ΟΗΕ για να διευκρινιστούν οι διαδικασίες, να δώσουμε οδηγίες στο προσωπικό, ούτως ώστε τα πάντα να βαίνουν ομαλώς. είναι σημαντικό να επιμείνουμε επί της καλής συνεργασίας. Θα ξέρετε ίσως ότι το ελεγκτικό συνέδριο παρέστη στην πρόσφατη ετήσια συνεδρίαση του φορέα που ελέγχει τον, το έργο της ΦΑΦΑ. Αυτό έγινε πέρσι στη Βιέννη. Και μετά από τη συζήτηση αυτή προσεκλήθη το ελεγχτικό συνέδριο να συναντήσει τους ομολόγους του στο σύστημα το ΙΕ. Έτσι θα βελτιωθεί συνεργασία στο μέλλον. Και εσείς Πρόεδρε αναφερθήκατε στο ενδιαφέρον της Κοκομπίου για το θέμα αυτό. Έγιναν εκτενείς συζητήσεις με την Επιτροπή Ενέχου Προπολογισμού και θα συζητήσουμε και με τον ΙΕ περαιτέρω την όλη λειτουργία του συστήματος. Δεν θέλω να σας δώσω αρνητική εικόνα για τη συνεργασία μας στον ΟΗΕ, κάτι που ίσως να βγαίνει από την αναφορά του ελεκτικού συνεδρίου. Βέβαια υπάρχουν προβλήματα και θα πρέπει να βρούμε τα αίτια των προβλημάτων αυτών. Και όπως υπογράμμισε ο εισηγητής θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη δέουσα πρόσβαση στα στοιχεία τους ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα χρήματα των φορολογουμένων χρησιμοποιούνται σωστά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ο Είναι σημαντικό να υπάρχει πλήρης κατανόηση του βασικού θέματος και συνεννόηση μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Νομίζω ότι πάνω σε αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε το, στη ζήτηση του σχεδίου γνωμοδοτήσεως Σεντιβάνη, κεφάλαιο 3, απαλλαγή 2007 και αν επιτρέπουν οι συγητές, εγώ θα προτείνω μια αλλαγή στην ημερήσια διάταξη. Θα πάμε παρεφής στο σημείο 16 της ημερήσιας διάταξης, ενδιάμεση αναθεώρηση του δημοσιονομικού πλαισίου 2007-2013. Αν δεν έχετε αντίρρηση, έχουν το σχέδιο γνωμοδοτήσεως του κύριου Μάικλ Γκάλερ. Σχέδιο γνωμοδότησης, δεν το έχετε στο φάκελο, αλλά διανεμήθη χωριστά. Ή το κείμενο υποστηρίζει την προσέγγιση που ακολούθησε ο κ. Μπέγκερ, εισηγητής Επιτροπής Προπολογισμών. Θα δώσω το λόγο στον εισηγητή σαν ετών σας πω ότι αυτό το σχέδιο γνωμοδοτήσεως σωστά προσδίδει μεγάλη σημασία στη χρηματοδότηση του κεφαλαίου 4 είναι βασικό θέμα αν ειδωθεί από την ε, σκοπιά της Επιτροπής μας των εξωτερικών υποθέσεων, διότι πάντα πιστεύουμε ότι υπάρχει υποχρηματοδότηση διαθωτική αυτού του κεφαλαίου και αυτό ετέθηκε χθε όταν η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ε, αναφέρθηκε στο θέμα. Αν θέλουμε να παίξουμε το ρόλο μας πλήρως, χρειάζονται διαθωτικές αλλαγές όσον αφορά τη χρηματοδότηση και εμένει ο συντάκτης του κειμένου. Κύριε Γκάλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, έχετε πει τα ουσιαστικά. Και εδώ το κύριο σύντημα είναι η χρηματοδότηση στο σημείο στην κατηγορία 4 των δημοσιονομικών προοπτικών και εδώ πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε ό,τι αφορά τις ε, προσαρμογές στο πολιετές πλαίσιο. Έχουμε βέβαια βαχυπρόθεσμες λύσεις τις οποίες μπορούμε να επιφέρουμε, αλλά συγχρόνως χρειαζόμαστε για την επόμενη περίοδο δημοσιονομικού προσανατολισμού και λύσεις που ξεπερνούν αυτή τη χρονική υποχρηματοδότηση αυτής της κατηγορίας και βλέπουμε επίσης την ανάγκη να δημιουργήσουμε και ένα μηχανισμό ευκαμψίας ο οποίος θα μας επιτρέπει να αντιδρούμε σε απρόβλεπτες καταστάσεις όπως η τωρινή κατάσταση που είδαμε με την καταστροφή της Γάζας θα πρέπει να δούμε πού θα βρούμε τα λεφτά. και θα πρέπει να αποφύγουμε την αποδυνάμωση της χρηματοδότησης για άλλα προγράμματα και άλλες πολιτικές στον τομέα των εξωτερικών πολιτικών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κάτι τέτοιο. Μία επίσης αναφορά στο εργαλείο για την πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αρκετά, αρκετοί πόροι για να αντιμετωπίσουμε μέσα στα πλαίσια της πολιτικής αυτής τους προσδοκόμενους εταίρους. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πολιτική για να εξασφαλίσει την ασφάλεια και την ευμάρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις στον τομέα της ασφάλειας τροφοδοσίας σε ενέργεια, εγώ ζητώ από την Κομισιόν να προβλέψει κατάλληλα μέσα για να μπορέσει να μειώσει την τροτότητά της σε ό,τι αφορά την ε, τροφοδοσία σε ενέργεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ακόμα ένα σημείο που αφορά ένα άλλο εργαλείο <clears throat> στην εξωτερική μας δράση και αυτό είναι το μέσο για την ανάπτυξη και συνεργασία. Πρέπει να κλείσουμε εδώ το χάσμα μεταξύ της θωρινής εστίασης που είναι πάνω στην ανάπτυξη και τους στόχους ανάπτυξης της χιλιετίας από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά την συνεργασία με χώρες μέσου εισοδήματος και χώρες οι οποίες βρίσκονται σε πιο υψηλό στάδιο ανάπτυξης ώστε να έχουμε πολιτικές ευρύτερες από απλώς πολιτικές που εμπίπτουν στο, στην κατηγορία της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε τέτοιου είδους πολιτικές σε χώρες όπως είναι η Βραζιλία ή άλλες χώρες μέσου εισοδήματος και αναδυόμενες χώρες της Ασίας βάσει αυτού του μέσου γιατί δεν θα είχε θεωρηθεί αυτό το πράγμα αποδεκτό μέσα στις προδιαγραφές αυτού του είδους αναπτυξιακής βοήθειας και επομένω εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Κομισιόν να προτείνει τις κατάλληλες τροποποίησεις ώστε στο επόμενο <clears throat> πλαίσιο δημοσιονομικό θα υπάρχει ένα επαρκές ε, ποσό, ένα, θα υπάρχουν επαρκή κονδύλια για τη χρηματοδότηση ενεργειών συνεργασία με χώρε μέσου εισοδήματο. Αυτέ ήταν οι κύριε προτάσει, τι οποίε θα ήθελα να φέρω από την πλευρά, να δώσω στην Επιτροπή Προπολογισμών. Σα ευχαριστώ, ο εισηγητή. Σα ευχαριστώ την προσοχή στην μεγάλη σπουδαιότητα τη δημοσιονομικής αυτής διάσταση των εξωτερικών ε, υποθέσεων βασικές μου του κ. Γκάλερ γιατί <clears throat> αυτό είναι ο λόγος που θα χρησιμοποιούμε όταν θέλουμε να τονίσουμε τη σπουδαιότητα να δοθεί σημασία στην εξωτερική πολιτική σε Σεντίβανη. Καταρχάς να συγχαρώ τον κύριο Γκάλερ για μια σημαντικότατη συνεισφορά του στην παρουσίαση που έκανε και στην γνωμοδότηση που παρουσίασε. Πιστεύω ότι Πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό. Καταρχάς υπάρχει συνένεση στην Επιτροπή ότι οι εξωτερικές σχέσεις υποχρηματοδοτούνται. Η μόνη αποδεκτή και πραγματική ουσιαστική λύση είναι σημαντική, ουσιαστική αλλαγή των κονδυλίων, βελτίωση των κονδυλίων ε, για την εξωτερική πολιτική. Δεδομένου των πολιετών ε, δημοσιονομικών προοπτικών μέχρι το 2013 δεν πιστεύουμε ότι αυτό βράχει πρόθεσμα, μπορεί να αλλάξει, αλλά μέσω πρόθεσμα πρέπει. Χρειαζόμαστε περισσότερα κονδύλια, αυτό είναι απλό, και νέα, νέους πόρους. Ακόμα και κατά τη δεύτερη φάση των δημοσιονομικών προοπτικών. Θα έπρεπε λοιπόν να απαιτήσουμε μια ουσιαστική ενδιάμεση αναθεώρηση. Το δεύτερο ζήτημα που εύγλωτα υπογράμμισε ο κύριος Γκάλετ είναι η ευελιξία. Η ευελιξία είναι βασικό στοιχείο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών. Δεν είναι δυνατόν να παραμείνουμε στην υφιστάμενη κατάσταση. Μη τα κονδύλια να, επιτρέπονται, να επιστρέφονται συγγνώμη, στα κράτη-μέλη. Υπάρχουν πολλές σημαντικές ευθύνες που μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε. Να χρηματοδοτήσουμε. Χρειαζόμαστε λοιπόν ευελιξία και εντός και ανάμεσα στις κατηγορίες. Κατόπιν, ένα, μια σημαντική προτεραιότητα είναι να εμβαθύνουμε την ε, σχέση μεταξύ των κατηγοριών και να τονιστεί αυτό και στην ενδιάμεση αναθεώρηση. Μια τελευταία παρατήρηση. Η εξωτερική δράση πρέπει να χρηματοδοτείται από κοινοτικά κονδύλια, από τον προπολογισμό της κοινότητας. Αυτός πρέπει να είναι ο κανόνας και μόνο κατ' εξαίρεση να υπάρχει χρηματοδότηση εκτός κρατών μελών. Αυτό θα πρέπει να είναι η καθοδηγητήρια γραμμή. Αν θέλουμε να μας παίρνουν στα σοβαρά και αν πιστεύουμε όντως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παίξει έναν ρόλο στην παγκόσμια σκηνή, πρέπει να δεχθούμε την αρχή αυτή. Πέραν όλων των άλλων υποστηρίζω το, την έκθεση και ελπίζω η Επιτροπή μας να αναβαθμίσει τις προσπάθειες για να υπάρξει μια ουσιαστική ενδιάμεση αναθεώρηση. Μας το υποσχέθηκαν, πρέπει να το απαιτήσουμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Άντριου Νταφ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Να ρωτήσω κάτι. Η ερώτησή μου αφορά την προσέγγιση που θα ακολουθήσουμε όσον αφορά την συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ταμείου εντός του προπολογισμού της Ενώσεως. Η συνθήκη, εάν τεθεί σε ισχύ, θα πρέπει να ενθαρρύνει, θα πρέπει να επιτρέπει τουλάχιστον την πλήρη συμπερίληψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης στον προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εφόσον η αναπτυξιακή χρηματοδότηση είναι βασικό εργαλείο για την εξωτερική πολιτική και την πολιτική ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα μπορούσαμε να εξφραστούμε εδώ στην Επιτροπή μας επί του θέματος χωρίς να μπαίνουμε στα χωράφια της Επιτροπής Ανάπτυξης. Θα ήθελα, θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η άποψη του κυρίου Γκάλερ σχετικά με αυτό το θέμα. Ο κύριος Γκάλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, πάνω σε κάτι που ο κ. Σαντιβάνη που είπε ότι καταρχήν θα πρέπει όλες εξωτερικές δράσεις να ενταχθούν στον προπολογισμό εννοείται και στατιωτικές αποστολές και το μηχανισμό Αθηνά κλπ. Αυτό θα μπορούσα να το υποστηρίξω με τα χαράς. Όμως έχω αμφιβολίες. Δεν ξέρω αν τα κράτη-μέλη θα το δεχθούν τώρα. Φαντάζομαι όμως ότι μέσω τροπολογίας θα μπορούσα ρητά να αναφέρω όλα αυτά τα τμήματα της de facto πολιτικής που ακολουθούμε που δεν εντάσσεται στον προϋπολογισμό. Δεν εντάσσονται στον προϋπολογισμό. Στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας θα μπορούσα να συμπεριλάβω πτυχές και όπως είπε Άντριου Νταφ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης θα μπορούσε να συμπεριληφθεί. Είμαι υπέρ του να συμπεριληφθεί στον προπολογισμό, ίσως θα δοθεί ευκαιρία να προσθεθεί σχετική αναφορά στο κείμενο. Με τα χαράς να κάνω αυτή την προσθήκη. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Άλλος συνάδελφος ο οποίος επιθυμεί να πάρει το λόγο δεν βλέπω. υπάρχει κάποιος. Ευχαριστώ τη συντάχτη τον κύριο Γκάλερ για την έξοχη αυτή γνωμοδότηση η οποία πραγματικά αντικατοπτρίζει τη φιλοσοφία της Επιτροπής μας στον τομέα αυτό του προπολογισμού. Εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση πάνω στο θέμα. Οι τροπολογίες μπορεί να υποβληθούν μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Και καταρχήν θα έπρεπε να πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η Τουρκία. Σχέδιο ψηφίσματος για την έκθεση πρόοδου της Τουρκίας, για την Τουρκία, τη συναδέλφου Ρία Όμεν Ρόιτεν Έχουμε κάποιο τεχνικό προβληματάκι διότι η συνάδελφός μας ψηφίζει, διεξάγεται ψηφοφορία επί της εκθέσεώς της στην Επιτροπή Απασχόλησης και θα πρέπει να καταφτάσει η συνάδελφος στις 10.30. Γι' αυτό το λόγο, μην έχοντας άλλη λύση, διακόπτουμε μέχρι τις 10.30. yeah. Καθίστε αγαπητοί συνάδελφοι, ξαναρχίζουμε τις εργασίες μας. Θα συνεχίσουμε με το σημείο 13. Δεν θεωρώ ότι είναι γρουσούζικο νούμερο. Το ψήφισμα για την έκθεση πρώτης Τουρκίας για το 2008. Δίνω αμέσως το λόγο στην εισηγήτριά μας, κυρία Όμεν Ρόιτεν. Πρόεδρε. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα, από σεβασμό προς την Ολλανδική γλώσσα. Επιτρέψτε μου πρόεδρε να ξεκινήσω ευχαριστώντας όλους σας για την σημαντική συνεισφορά που προσφέρεται για την υλοποίηση της έκθεσης. Οι περισσότερες τροπολογίες που έχουν υποβληθεί είναι επικοδομητικές και ξεκίνησε τις συζητήσεις με τους σκιώδεις συζητητές ακριβώς κάτω από αυτή την οπτική γωνία. Έχω υποβάλει 13 συμβαστικές προτάσεις τροπολογίες ενώ θα προσθεθούν και κάποιες προφορικές τροπολογίες. Εισαγωγικά να προσθέσω τα εξής φέτος είχαμε λιγότερες τροπολογίες από πέρυσι. Πιστεύω ότι εν γέννη συμφωνούν όλοι με τις προτεραιότητες που αναφέρω στην πρώτη, στις πρώτες παραγράφου. Είχα τονίσει εκεί ότι υπάρχουν τέσσερα βασικά σημεία. Λίγα πράγματα έγιναν σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις κατά το 2008. Πρέπει λοιπόν να επιταχυνθεί ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων. Και οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις ιδιαίτερες, δηλαδή τα κριτήρια της Κοπενχάγης, αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Τέταρτο σημείο, η πόλωση στην τουρκική πολιτική σκηνή και την τουρκική κοινωνία αποτελεί κάτι κακό για την διαδικασία μεταρρυθμίσεων. Στην έκθεσή μου υπογράμμισα αυτά τα τέσσερα σημεία. Πρώτον, στήριση των κριτηρίων της Κοπενχάγης, αύξηση του επίπεδου ευημερία, ενίσχυση της ευημερία, θέσπιση σχέσεων, οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας και ενίσχυση των διμερών συνεργασιών. Ε, εμένοντας και υπογραμμίζοντας τα κριτήρια της Κοπενχάγης, ε, πέραν μάλλον των κριτηρίων της Κοπεχάγης, πιστεύω ότι η ενίσχυση της ευημερίας και της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής στην κοινωνία αποτελούν κάτι πολύ σημαντικό και για την Τουρκία βεβαίω, αλλά και για μας. Επίσης, θέλω να ζητήσω να υπάρξει καλύτερη προστασία και μεγαλύτερη και περισσότερα δικαιώματα για όλες τις θρησκευτικέ κοινότητες. Συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, δεν ανοίγουμε κεφάλαια, δεν είναι αυτό το βασικό ζήτημα. Ο στόχος είναι να συνεχίσουμε τον εξυγχρονισμό και τον εκδημοκρατισμό της τουρκικής κοινωνίας. Θα ήθελα, Πρόεδρε, να ασχοληθώ με τις τροπολογίες. Όπως είπα, κάποιες προτάσεις συναδέλφων τις υιοθέτησα. Σε κάποια άλλα κείμενα υπήρχαν συμβιβασμοί με τους σκιώδεις εισηγητές. Κάποιες τοπολογίες δεν τις δέχτηκα γιατί όχι μόνο θα γινόταν ε, χριστουγεννιάτικο δέντρο η έκθεση, αλλά διότι θα χανόντουσαν και τα μηνύματα που θέλουμε να δώσουμε αν κάθε φορά επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια. Σε ό,τι αφορά την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης, καθώς και την καταπολέμηση των διακρίσεων, των, την υποστήριξη των δικαιωμάτων των γυναικών, τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών και των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, τα συμβιβασ... οι συμβιβασμοί είναι ξεκάθαροι συμφωνήσαμε. Ζητώ λοιπόν την υποστήριξη των συναδέλφων για τις προτάσεις αυτές και ευχαριστώ τους και ηγητές για τον τρόπο με τον οποίο συνέβαλαν στην υλοποίηση της έκθεσης αυτής. Όπως είπα κάποιες άλλες τροπολογίες θα ζητούσα να τις καταψηφίσουμε πρόεδρε. Το ψήφισμα ασχολείται με την εξέλιξη της Τουρκίας το 2008. Δεν πρέπει να επαναφέρουμε στοιχεία ε, που δεν σχετίζονται με την κατάσταση. Ο κύριος Χάουιτ έκανε μια σειρά προτάσεων, τροπολογία 36. Ε, για την τροπολογία 36 είχα συζητήσει με τον κύριο Βίσμα και τον κύριο Σβόμποντα. Ε, πήραμε και κάποιες πληροφορίες από την Επιτροπή. Το θέμα είναι η συνεπροτοχή του ΔΤΠ στην εκλογική επιτροπή. Ε, τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξα είναι ότι η τροπολογία αυτή δεν ήταν ακριβής, δεν ήταν σωστή. Θα μπορούσαμε μέχρι την Ολομέλεια να βρούμε μια άλλη διατύπωση, αλλά το κείμενο έχει τώρα, δεν με βρίσκει σύμφωνη και ζητώ την καταψήφισή του. Ζητώ από τον Χάνες να αποσύρει αν γίνεται η τροπολογία αυτή. Κατόπιν, παράγραφος 38, δική μου. Και εδώ υπήρχαν κάποιες παρατηρήσεις και σχόλια. Πιστεύω ότι το Belli δεν, η απόσυρση του Κάσου Belli δεν, δεν είναι καθόλου προβληματικό. Πιστεύω ότι η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μέσα στο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Ε, μετά, για την Τελωνιακή Ένωση. Χαίρο διότι ο Υπουργό Εξωτερικών στις 8 Δεκεμβρίου του 8 δήλωσε ο, σαφέστατα ότι επήγει να υπάρξει πρόοδος. Το 2006 το Συμβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή για την περίοδο 2007, 2008 και 2009 να υπάρχουν εκθέσεις σχετικά. Το 2009 ε, η απόφαση δηλαδή το 2009 προκύπτει από, δεν θα ισχύσει γιατί ε, αυτό προκύπτει από την απόφαση του Συμβουλίου της 11 Δεκεμβρίου του 2006. Το υπογραμμίζω αυτό. Δεν ε, καταργούμε εμείς την ημερομηνία 2009. Η ίδια η Τουρκία πρέπει να κάνει τη δουλειά που πρέπει να υλοποιηθεί μέχρι το 2000, που έπρεπε να υλοποιηθεί μέχρι το 2009. Οι συνάδελφοι που θέλουν να καταργηθεί η ημερομηνία αυτή θα πρέπει να το ξανασκεφτούν. Επίσης, πρόεδρε, η εξέλιξη, η εξέλιξη στην ίδια την Τουρκία τώρα. Ίσως να υπερτιμώ τον ρόλο μας στο σημείο αυτό. Με την έκθεση πρόοδου της Επιτροπής ωστόσο και την επίσκεψη της, Επιτροπ... της αντιπροσωπείας μας στην Άγκυρα, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 8 η Δεκεμβρίου και την πρώτη συζήτηση που είχαμε για την έκθεση με οδηγούν όλα αυτά στο να έχω την εντύπωση ότι το μήνυμα περνά, πέρασε στην Τουρκία. Γιατί τώρα υπάρχει ένα εθνικό πρόγραμμα για την ενσωμάτωση του κεκτημένου και ένας νέος διαπραγματευτής, ο κ. Μπαγκής, ο οποίος εργάζεται full time για το θέμα της ευρωπαϊκής προσχώρησης. Ένα σημαντικό ζήτημα. Χτες συζήτησα με τον κύριο Μπαγκής, μιλήσαμε επί μακρόν για την έκθεση. Οι εκπομπές τηλεοπτικών σταθμών στα κουρδικά και οι συγκεκριμένες επαφές της κυβέρνησης με τους αλεβίτες αποτελούν καλό μήνυμα που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Είναι λυπηρό ωστόσο ότι δεν έχουμε μόνο καλά νέα. Ο νόμος για τον διαμεσολαβητή ακυρώθηκε από το συνταγματικό δικαστήριο παρά την καλή εντύπωση που ε, μας είχε κάνει ο κύριος Ερντογκάν να αναφέρθηκε στο σημείο αυτό όταν είχε έρθει στις Βρυξέλλες πριν από 2-3 εβδομάδες. Παρά τα αυτά έχουμε κάποια ερωτήματα, ιδιαίτερα για το σχέδιο Ναμπούκο. Για να σας πω την αλήθεια πρόεδρε, θα ήθελα όταν, την, όταν ψηφίσουμε την έκθεση να αποτελέσει το αποτέλεσμα ένα κίνητρο, μια παρότερη προς την Τουρκία, ούτως ώστε να αναλάβει τις ευθύνες της. Ως κοινοβούλιο πρέπει να περάσουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να πούμε ότι οι μεταρρυθμίσεις είναι αναγκαίες για την Τουρκία, ούτως ώστε να μπορέσει η χώρα αυτή να αναπτυχθεί και να γίνει ένα σύγχρονο κράτος με μια κοινωνία που θα γνωρίζει την κοινωνική ευημερία. Προς την κατεύθυνση αυτή θέλουμε με υπεύθυνο τρόπο να συμβάλλουμε. Ελπίζω ότι θα έχουμε ε, ευρεία ε, πλειοψηφία στην έγκριση της έκθεσης όπως και την προηγούμενη φορά και ελπίζω ότι αυτό θα περάσει καλύτερα τα πράγματα. Σας ευχαριστώ. Thank you well. Ευχαριστώ πολύ, λέει και ο Πρόεδρος. Θα δώσω το λόγο στους κοιόδης εισηγητές γιατί έχουμε και περιορισμό χρόνου. Δυόμιση λεπτά στον καθένα σας παρακαλώ. Ο Χάνες Φόμποντα, ο οποίος είναι ο σκιώδης ηγητής για τους σοσιαλιστές και ήταν και ο επικεφαλής αντιπροσωπείας που πήγε τον Νοέμβριο στην Άγκυρα, ο Χάνες. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να σύντομεύσω όσο μπορώ. Θέλω να πω σαφώς ότι θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας στην ε, Ρία για την πολύ καλή έκθεσή της και την πολύ καλή συνεργασία της με τους σκιώδεις εισηγητές. Εγώ πράγματι ως ε, επικεφαλής αντιπροσωπείας στην Τουρκία μπορώ να πω ότι είχαμε επαφές με τον πρόεδρο, τον ε, Πρωθυπουργό τη Τουρκία μα δέχτηκαν με μεγάλο σεβασμό και ενδιαφέρον και ήταν πολύ θετικά τα, στι, τα μηνύματα από την Τουρκία. Βέβαια υπάρχουν και ρεύματα τα οποία θέλουν να τροχοπεδίσουν την διαδικασία μεταρρύθμιση στην Τουρκία και επομένω η έκθεση τη ΡΙΑ δίνει δύο μηνύματα. Καταρχήν υπάρχει το θετικό μήνυμα για τα πράγματα τα οποία πηγαίνουν θετικά, αλλά υπάρχουν και από την άλλη πλευρά σημεία στα οποία έχουν τελματώσει τα πράγματα και εκεί εμεί θα πρέπει να ασκήσουμε κάποια πίεση. Οι συμβαστικέ τροπολογίε, οι οποίε έχουν τύχει διαπραγμάτευση είναι πολύ θετικέ. μπορώ να τι συνιστήσω, να τι υποστηρίξουν, να τις υποστηρίξουν οι συνάδελφοι. Και για τα δύο σημεία τώρα που ανέφερε η συγκήτρια για την τροπολογία 36. Καταρχήν αυτό το οποίο λέει είναι σωστό, ότι τα κόμματα τα οποία τώρα ε, είναι υποψήφια σε εκλογές, αλλά δεν ήταν μέσα στην εκλογική διαδικασία στις προηγούμενες εκλογές δεν έχουν κανένα δικαίωμα να είναι παρόντα στην ελεκτική εκλογική επιτροπή στα συγκεκριμένα εκλογικά τμήματα να εκπροσωπούνται. Αυτό είναι βέβαια άδικο, αλλά είναι δύσκολο να το τροποποιήσουμε τώρα. Καταρχήν όμως είναι σωστό να παραμείνουμε λοιπόν, να, θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω να ανατροποποιηθεί αυτή η, η τροπολογία και να έχουμε ένα κοινό ψήφισμα, μια κοινή τροπολογία μάλλον η οποία θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο αυτό θέμα. Να πούμε λοιπόν στην τροπολογία αυτή ότι στο μέλλον θα πρέπει να υπάρχει μια νομική διευκρίνηση η οποία λέει ότι όλοι οι υποψήφοι το, όλα τα υποψήφια κόμματα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην εκλογική επιτροπή. Αυτό είναι λοιπόν κάτι το οποίο εγώ θα υποστηρίξω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πρόβλημα για κάτι τέτοιο. Το, το πρόβλημα επίσης που είναι δύσκολο είναι το θέμα για την καταληκτική ημερομηνία του 2009. Υπάρχουν τροπολογίες οι οποίες επιτείνουν αυτή την καταληκτική προθεσμία, άλλες τροπολογίες θέλουν να υπάρχει χαλάρωσή της. Αυτό που δεν θέλει η πολιτική ομάδα είναι να υπάρξει ένας αυτοματισμός, δηλαδή αν περάσει το 2009 χωρίς κάποια πρόοδο, να υπάρξει αυτοματισμός ότι εμείς δεν θα προχωρήσουμε στις διαπραγματεύσεις με την Τουρκία θα τροχοπεριθούν, θα σταματήσουν αυτομάτως οι διαπραγματεύσεις. Αυτό νομίζω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί μηχανιστικά. Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολιτικό θέμα εκτίμησης. Εγώ μπορώ να φανταστώ ότι μπορούμε να δεχτούμε καταρχήν το κείμενο της ΡΙΑ όταν έχουμε πει επιπλέον όμως ότι δεν θα πρέπει να υπάρξει μια μηχανιστική, αυτοματιστική διαδικασία που θα οδηγήσει στην απόλυτη τροχοπέδηση των διαπραγματεύσεων. Μπορούμε να συζητήσουμε τώρα κατά πόσο μπορούμε να συζητήσουμε με τους συναδέλφους αν μπορούν να δεχτούν το κείμενο αυτό συμβιβαστικό με την ΡΙΑ και μπορώ το απόγευμα να κάνω συνεννοήσεις με την πολιτική μου ομάδα και να σας πω μετά κατά πόσο μπορούμε να αποδεχτούμε αυτή τη συμβιβαστική λύση. Παρακαλώ λοιπόν να είσαστε μέσα στον χρόνο ο Άντριου Ντάφ για τους φιλελεύθερους. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την θαυμάσια έκθεσή της, η οποία έχει αποκομίσει και μια ευρεία συνένεση χάρη στη συνενετική τακτική που ακολούθησε η συγγήτρια. Εμείς υποστηρίζουμε αυτή την έκθεση, θεωρούμε ότι είναι αρκετά επιφυλακτική και έχει και το σωστό κριτικό πνεύμα. Παρόλα αυτά είναι μια έκθεση η οποία έχει ενθαρρυντικό χαρακτήρα προς την Τουρκία, την ενθαρρύνει να συνεχίσει την διαδικασία ένταξη στην πορεία προς την ένταξη και τις μεταρρυθμίσεις. Θα πρέπει να δεχτούμε όλοι ότι υπάρχουν δύο θέματα τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν, αλλά δεν είναι ακόμα σε θέση να αξιολογήσουν πλήρως αυτά τα στοιχεία. Το πρώτο είναι ο αντίκτυπος οικονομικής κρίσης στην Τουρκία, που νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ενδεχομένως θα φτάσει ένα επίπεδο που θα είναι ανάλογο αυτό σε άλλες αυτού σε άλλες χώρες αλλά βλέπουμε ότι μπορεί να υπάρξει και μια κατάρρευση του εμπορικού ισοζυγίου της Τουρκίας και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το αποκλείσουμε, θα πρέπει να το προβλέψουμε. Το δεύτερο θέμα στο οποίο όπου δεν μπορούμε να εκφέρουμε γνώ, γνώμη με μεγάλη ασφάλεια είναι το σκάνδαλο του Εργενεκών. Σίγουρα είναι μια σκανδαλώδης κατάσταση. Αλλά πιο σημαντικό είναι να κατανοήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει και να δούμε ποια στοιχεία μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποτελούν μια απλώς εγκληματική ε, δραστηριότητα και ποια είναι απλώς πολιτική εκμετάλλευση. Και εγώ συμμερίζομαι την λύπη της εισηγήτριας ότι οι εντάσεις μεταξύ της κοσμικής και της θρησκευτική πτέρυγας στην Τουρκία φαίνεται να ενισχύονται όπως και οι εντάσεις μεταξύ του στρατού και του ΑΚΠ. Επίσης η ημερομηνία του 2009 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη με κατανόηση σε ό,τι αφορά την κατάσταση στην Τουρκία. Επίσης για τις συμβιβαστικές τροπολογίες. Η τροπολογία 12 για την Κύπρο. Η Κύπρος αποτελεί μια προτεραιότητα, η λύση του Κυπριακού αποτελεί μια προτεραιότητα για όλους μας σε αυτό το 12 διάστημα. Πιστεύω ότι υπάρχει μια ευκαιρία για τους κυρίους Ταλάτ και Χριστόφια να επιτύχουν μια πραγματικά ιστορική ρίξει με το παρελθόν και μία λύση για την Κύπρο. Ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βοηθήσει αυτή τη διαδικασία περισσότερο και αυτό θα επιτευχθεί αν μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο κλίμα μέσα στο οποίο μπορούν να λάβουν χώρα οι διαπραγματεύσεις. Και σε αυτό θα ευνο... στις διαπραγματεύσεις θα είναι πολύ θετικό αν η Τουρκία αποσύρει τα στρατεύματά της ή το μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον των στρατευμάτων της από την Βόρεια Κύπρο γιατί δεν είναι πραγματιστικό ούτε εφικτό να αναμένουμε μια πλήρη αποχώρηση στρατευμάτων προτού επιτευχθεί μια πλήρης και οριστική λύση για το Κυπριακό και να μπορέσει να υπερνικηθεί η ιέρε του νησιού. Ευχαριστώ. Ο Σιμάνσκι, λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ καλή η έκθεση. Προφανώς έχουμε μια πολύ ισορροπημένη προσέγγιση ως προς τις εσωτερικές ε, πολιτικές της Τουρκίας και ως προς τις εξωτερικές σχέσεις της Τουρκίας με τους γείτονές της ε, έχουμε επισημάνει τα βασικά σημεία, κυρίως την ενεργειακή πολιτική. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιατί αναφέρεστε και στις ε, θρησκευτικές ελευθερίες. Κάτι τέτοιο δεν θα μπορούσε να είχε γίνει χωρίς πιέσεις από την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ουσιαστική πρόεδρος προς αυτή την κατεύθυνση και ε, θεωρούμε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να βελτιωθεί και να εφαρμοστεί. Μας ενδιαφέρουν τα θέματα των επιστροφών περιουσιών, την ε, ε, δυνατότητα να διδάσκουν ιερείς και ε, εγώ ξέρω πάρα πολύ καλά ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν πριν προετοιμάσουμε την ένταξη της Τουρκίας. Είμαι ο τελευταίος ίσως εδώ που θα μπορούσε να μιλάει για θέματα θρησκευτικής ελευθερίας, αλλά οι θρησκευτικές ελευθερίες είναι στην καρδιά των αξιών μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στη διεθνή αρένα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μπορούμε πάντα να αναφερθούμε για τα, στα θέματα αυτά στην έκθεσή μας. Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαμε να αναφερθούμε και σε κάποια θέματα ως προς την ε, πιο ήπια νομοθεσία. Παραδείγματο χάρη για την ε, προστασία των ε, σεξουαλικών νομο... μειονοτήτων στην Συμβαστική Τροπολογία 5. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω καταρχάς την εισηγήτρια για τον τρόπο με τον οποίο προσπαθήσε να βρει μια συμβιβαστική λύση στις τροπολογίες η ομάδα μου θα υποστηρίξει την πλειονότητά τους, διότι θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ καλές. Να σας δώσω τρία παραδείγματα. Αντίθετα με αυτά που λέει ο κ. Σιμάνσκι, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένο με τη συμβιβαστική τροπολογία 5 ε, που υποστηρίζει την Λάμδα Ινσταμπούλ, μια οργάνωση που προσπίζει τα δικαιώματα των ε, ομοφιλοφίλων. Επίσης, Χαίρομαι για την τροπολογία που αναφέρεται στην δυνατότητα που έχουμε να ε, επικοινωνούν οι πολίτες στα κουρδικά στην ε, περιφέρειά τους. Υπάρχει ε, πλέον και το κανάλι ε, το κουρδικό το οποίο λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο και επίσης με χαροποιεί και η τροπολογία 11 που υποστηρίζει τις δυνατότητες που έχει το κουρδικό κοινοβούλιο να ξεκινήσει τις εργασίες του και επίσης επιβάλλει στην κυβέρνηση να βρει μια λύση για το θέμα των ε, διαδηλώσεων. Δεν μου αρέσουν οι τροπολογίες 10 που επιτρέπουν την, ε, τις ε, συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου με τρίτες χώρες και αποκλείεται η Τουρκία. Ε, ίσως ε, θα έπρεπε να αναφερθεί στο μέλλον, να συμπεριληφθεί η Τουρκία, ίσως να πηγαίνουμε λίγο παραπέρα από θα ήθελε η, η, η εισηγήτρια. Ίσως θα μπορούσαμε να αλλάξουμε λίγο τη διατύπωση και να λέμε να διαβουλευόμαστε την Τουρκία για αυτές τις συμφωνίες. Ε, εκείνη η τροπολογία βέβαια που δεν μου αρέσει καθόλου είναι το θέμα της Κύπρου και των θεμελιωδών δευτεριών. Φαίνεται πάρα πολύ λογικό να το κάνουν οι Ευρωβουλευτές και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά δεν είναι σωστό. Η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι τούδε ήταν να δεχόμαστε παρεκκλήσεις ε, από τις τέσσερις ελευθερίες που είναι τμήμα του κοινωτικού κεκτημένου, έστω και προσωρινά. Η πρόταση Ανάντ, την οποία είχε χαιρετήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περιείχε προσωρινέ παρεκκλήσει για τι τέσσερι ελευθερίε. Γιατί να αλλάξουμε αυτή τη θέση όμω τώρα. Είναι μια θέση την οποία έχει δεχτεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο παρελθόν και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ προτείνω λοιπόν να μείνουμε στην άγουσα που είχαμε πάντα υποστηρίξει, διότι είμαι πεπισμένο ότι αυτή τη στιγμή ξαφνικά αναφερόμαστε στι τέσσερι ελευθερίε και αυτό σημαίνει ότι υπονομεύουμε τι δυνατότητε τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και του Συμβουλίου να κάνει οποιαδήποτε συμφωνία συμφωνία μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Ε, αυτό είναι αυτό που ίσως θα ήθελα να έχουν οι Ελληνοκύπροι συνάδελφοι, αλλά δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε τους Κιώδης, τα τακτικά μέλη, ο κύριος Δημητρακόπουλος. Και ο καθένας από εσά θα έχει δύο λεπτά, κύριε Δημητρακόπουλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν ε, θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Όμεν για την εργασία την οποία παρουσίασε όπως επίσης και για τις προσπάθειες τις οποίες ε, έκανε έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε μια ε, συμβιβαστική και κοινά αποδεκτή θέση. Έχω τρία σημεία πάρα πολύ γρήγορα. Το πρώτο σημείο για να ξεκινήσω από τα ευρωπαϊκά και να κατέβω στα περιοχικά. Το πρώτο σημείο αφορά τα θέματα της ενέργειας όπου θεωρώ ότι επειδή είναι πολύ σοβαρά ζητήματα πρέπει βεβαίως και εμείς να είμαστε προσεκτικοί αλλά πρέπει και η Τουρκία να είναι προσεκτική στα θέματα της ενέργειας και δεν νομίζω ότι εξάρσεις όπως η τελευταία σχετικά με μία πτυχή της ενέργειας γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Ναμπούκο είναι μία πτυχή της ενέργειας υπάρχουν και άλλες ε, δεν βοηθούν το δεύτερο σημείο είναι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις μειονότητες. Και το ξέρουμε και το έχουμε πει ότι η Τουρκία πρέπει να κάνει, έχει πολλά βήματα ακόμα να κάνει, σε ό,τι αφορά τον πλήρη και απόλυτο σεβασμό των δικαιωμάτων των μειονοτήτων και σε αυτή την κατεύθυνση η κυρία Όμεν πράγματι έχει πολύ σημαντικές ε, προτάσεις. Το τρίτο αφορά στο ζήτημα του Κάζους Μπέλη. Χαίρομαι ειλικρινά γιατί η κυρία Όμεν επιμένει σωστά κατά την άποψή μου στην αρχική της θέση ότι το κάζους Μπέλη πρέπει να αρθεί μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Στον 21ο αιώνα τέτοιου τύπου απειλές οπωσδήποτε δεν συμβαδίζουν με την ευρωπαϊκή προπτική μιας χώρας την οποία ευρωπαϊκή προπτική της Τουρκίας στηρίζουμε. Έτσι, το ξεκαθαρίζω αυτό. Τέλος, σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, και τελειώνω με αυτό, άκουσα και κάποια πράγματα βεβαίως σεβαστά ως απόψεις σχετικά με τις τέσσερες ελευθερίες και τα ζητήματα που είχε το σχέδιο Ανάν και τούτο και εκείνο και τ' άλλο. Εγώ θεωρώ ότι η διατύπωση που μιλάει για την αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων έτσι ώστε να διευκολυνθεί η σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Χριστόφιας με τον Ταλάτ είναι σημαντική θέση και δεύτερον δεν θα ήθελα να ξαναφέρουμε στην αίθουσα αυτή το σχέδιο Ανάν διότι το σχέδιο Ανάν έχει πεθάνει. Ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ο κ. Έγκερ είναι ο επόμενος. Thank you. <clears throat> Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρο και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Ρία η οποία έκανε τεράστια προσπάθεια για να μπορέσει να καταλήξει σε μια ισορροπημένη έκθεση. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου εύκολο για να εισηγητή μια έκθεση για την Τουρκία να καταλήξει σε συμβαστικέ θέσει. Γιατί υπάρχουν και οι υπέρμαχοι και οι αντίπαλοι τη ένταξη τη Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση όπω ξέρουμε όλοι. Τώρα θα ήθελα να πω το εξή, ότι είναι πλήρη φυσικά η έκθεση τη κυρία Φων Θέλω να σταθώ σε τρία σημεία. Έχω καταθέσει πάνω από 30 τροπολογίες με πολλούς συναδέλφους, τώρα κάποιες από αυτές τις τροπολογίες θα αποσύρθουν. Εγώ λέω στην, θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω την τροπολογία 41 που λέμε ότι τόσο η Τουρκία όσο και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεχίσουν τη δυναμική ένταξη και να την ενισχύσουν και αυτό να γίνει επί τη βάση ενός επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των δύο ε, εταίρων και για την υποστήριξη του δημόσιου διαλόγου στην Τουρκία για τα θέματα αυτά. Ξέρουμε ότι έχουν αναδυθεί προβλήματα στην Τουρκία και επίσης αυτά οφείλονται στη θέση ορισμένων Ευρωπαίων πολιτικών που δεν έκανε τους Τούρκους να νιώθουν ιδιαίτερα καλό στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα συγκεκριμένο επίσης θέμα είναι η Τελωνιακή Ένωση. Υπάρχει το θέμα της στήριξης των υποχρεώσεων της Τουρκίας έναντι της Τελωνιακής Ένωσης. Ναι, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχαν πολλές υποχρεώσεις οι οποίες δεν έχουν τηρηθεί. Εξακολουθούν να υπάρχουν περιορισμοί για τα τουρκικά φορτηγά προς την Ευρώπη. Μόνο το 1 τέταρτο των καμιονιών από την Τουρκία περνούν από ό,τι στο παρελθόν. Και αυτό θα πρέπει να το αναφέρουμε λοιπόν ότι υπάρχουν και από την πλευρά της Ευρώπης περιορισμοί στα πλαίσια της Θελωνιακής Ένωσης. Δεν πρέπει να παρουσιάσετε μονάχα ότι δεν έχει τηρηθεί το σύνολο των υποχρεώσεων από την πλευρά της Τουρκίας. Τέλος. Το τέλος του 2009 ως καταληκτική ημερομηνία, αλλά τι θέλουμε να πετύχουμε. Είπε η Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριος της ε, Γερμανίας, ότι ήταν εσφάλμα το να δεχτούμε την Τουρκία μονομερός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρουμε λοιπόν ότι εάν κρατήσουμε αυτή την ημερομηνία το 2009 σαν καταληκτική ημερομηνία, αυτό θα είναι λάθος απέναντι στην Τουρκία. Θα πρέπει να κάνουμε μια έκκληση και από τις δύο πλευρές να γίνουν οι απαραίτητες προσπάθειες για να επιληθεί το πρόβλημα αυτό το οποίο ισχύει. Δεν μπορεί η Τουρκία από μόνη της να λύσει τα προβλήματα αυτά. Θέλουμε η Τουρκία να είναι εταίρος μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να θέσουμε και δεν μπορούμε να θέσουμε λοιπόν σαν προϋπόθεση ότι θα υπάρξει επανένωση της, της Κύπρου πρωτού φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Ο κ. Ματσάκης. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Αμέν Ράιτεν για την έξοχη έκθεσή της για μία ακόμη φορά. Είναι έξοχη έκθεση και κατέβαλε μεγάλες προσπάθειες όχι μόνο για την έκθεση αλλά επίσης για τις συμβαστικές τροπολογίες. Πραγματικά αξιοσημείωτη η δουλειά της διότι επέφερε ισορροπία αλλά επίσης ήταν και ακριβωδίκαιη, κάτι που είναι απαραίτητο σε αυτή τη φάση. Διότι κύριε Πρόεδρε, αυτό που είδαμε τα τελευταία χρόνια ήταν το εξή. Αυτέ οι εκθέσει μετατρέπονται σε εκθέσει μη πρόοδου τη Τουρκία, Διότι η Τουρκία δεν σημειώνει την δέουσα πρόοδο και δίναμε στην Τουρκία αρκετά καρότα αυτά τα χρόνια και είναι και η ώρα να χρησιμοποιήσουμε και λίγο και το ραβδί. Το είπα την προηγούμενη φορά, την περασμένη εβδομάδα και πέρσι τα είχα πει και φοβάμαι ότι ισχύει και φέτος. Και είχαμε το παράδειγμα, δύο παραδείγματα που θα θέλω να παραθέσω. Ένα παράδειγμα είναι η παρουσία του τουρκικού στρατού κατοχή σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εξακολουθεί να είναι εκεί. Έχουμε 45.000 Τουρκικού. Τούρκους στρατιώτες που κατέχουν ένα κομμάτι κράτους μέλους. Και πώς μπορεί κανείς να πει ότι οι Τουρκοκύπροι ζητούν την προστασία του τουρκικού στρατού όταν οι Τουρκοκύπροι είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσέχει τους πολίτες τα τελευταία 50 χρόνια και προστάτευε την ευμάρειά τους και την ασφάλειά τους, την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών τα τελευταία 50 χρόνια. Τα τουρκικά στατεύματα κατοχής λοιπόν δεν χρειάζονται στην Κύπρο και νομίζω ότι εξαρτάται από την τουρκική κυβέρνηση να το κατανοήσει αυτό και να αποσύρει τα στατεύματα αυτά από την Κύπρο. Είναι απόφαση του Συμβουλίου η προθεσμία του 2009, συμπεριλαμβάνεται στην έκθεση Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπήρξαμε διπλωματικοί, υπήρξαμε, ήμασταν ανεκτικοί, καλοί, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε την Τουρκία επί πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι και, και η ώρα να θέσουμε μια προθεσμία. Θα πρέπει να κάνουν κάτι θα πρέπει να αρχίσουν να συμπεριφέρονται με ευρωπαϊκό τρόπο. Όχι για δικό μας όφελος, αλλά για δικό τους όφελος, για όφελος του λαού τους. Διότι εμείς θέλουμε να συμβούν αλλαγές στην Τουρκία. Εγώ θα έλεγα ότι η προθεσμία του 2009 πρέπει να τηρηθεί και τα τουρκικά στατεύματα κατοχής θα πρέπει να αποχωρήσουν από την Κύπρο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ματσάκη. Ο κύριος Μάτης έχει το λόγο. Μάτσης. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα με τη σειρά μου να εκφράσω την ικανοποίησή μας διότι η έκθεση της κυρίας Σόιμα σε έναν πολύ δύσκολο θέμα είναι αξιοπρόσεκτη, είναι σοβαρή και την υιοθετούμε χωρίς καμία επιφύλαξη. Θα ήθελα να τονίσω ότι σαν Κύπριος βουλευτής εσθεναρός και μόνιμα υποστηρίζω την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρώπη. Θα ήθελα όμως να τονίσω ότι αυτή η ένταξη με τα πολλαπλά προβλήματα που υπάρχουν εσωτερικά στην Τουρκία αλλά και με το Κυπριακό πρέπει να οδηγήσει τους ηθήνοντες στην Τουρκία να πάρουν τις σωστές αποφάσεις προσαρμογής με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Θέλω να τονίσω δύο σημεία για να μην μπω στα πολλά σημεία που τονίσαμε κατά επανάληψη. Πρόσφατα έχει αποκαλυφθεί ότι με χρηματοδότηση της ίδιας της Τουρκίας αγοράζονται και αξιοποιούνται τεράστιες εκτάσεις γης στην κατεχόμενη Κύπρο και ιδιαίτερα στην Καρπασία αλλά και παντού και αυτό παραβιάζει μία από τις σοβαρότερες αρχές που υποστηρίζεται και υιοθετείται στην Ευρώπη. Μία από τις τέσσερις βασικές αρχές. Γι' αυτό θέλω να διαφωνήσω με τον φίλο κύριο Λάγκερτα ότι πρέπει να δείξουμε ε, επιφυλακτικότητα σε αυτές τις θέσεις. Στο τέλος θα οδηγηθούμε σε μια κατάσταση ανεπίστρεπτη και δεν θα μπορούμε να λύσουμε το Κυπριακό με βάση των συμφέρων των Τουρκοκυπρίων και των Ελληνοκυπρίων. Δεν θα αναφερθώ την πρόσφατον θλιβερό γεγονός που απεκαλύφθη από τηλεοράσεως της εκτέλεσης από Τούρκο στρατιώτη 10 ε, κρατουμένων Ελληνοκυπρίων. Απλώς ήθελα να καταλήξω λέγοντας ότι το σχέδιο να έπαυσε να εφίσταται κατεψηφίστη από το 76% των Ελληνοκυπρίων και από το 36% των Τουρκοκυπρίων οι οποίοι σε αναλογία είναι όσοι περίπου το κατεψήφισαν και οι Ελληνοκύπροι διότι εψήφισαν οι περισσότεροι έπικοι υπέρ του σχεδίου. Οι Τουρκοκύπροι σε ποσοστό 36% το κατεψήφισαν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κ. Πριμπέτιτς. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για την σύνθετη και δύσκολη δουλειά που διεξήγαγε για την ενδιάμεση έκθεση και να σας πω τη δική μου άποψη την ανάγκη να υπάρξει ένα σαφές μήνυμα που θα στηρίζεται στην εξέλιξη της Τουρκίας και τον σεβασμό αυτών των στοιχείων κριτήρια της Κοπενχάγης, ευημερία, καλές σχέσεις, καλές γειτονίες και ενίσχυση της δημιουργού συνεργασίας. Να τονίσω δύο θέματα που ε, τόνισε και ο κύριος Βόμποντα. Την αναγκαιότητα να υπάρξουν συμβιβαστικές τροπολογίες, ειδικότερα να επανέλθει ένα δυνατό σημείο για την ε, τελ, τελειωτική μεμνία του 2009. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε μία ημερομηνία, μία διπλωματική θέση, να αφήσουμε στην ημερομηνία ευελιξία ωστόσο για να μην μπέσουμε σε, έναν, ε, σε μια μηχανική αντιμετώπιση της κατάστασης με μια σειρά συνεπειών που θα μας απομάκρυνε από τον δρόμο που θέλουμε να ακολουθήσουμε για την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Δεύτερο θέμα, σύντομα. Το σημείο 37 όπου εκφράζουμε την ικανοποίησή μας για την πρόοδο ό,τι αφορά την, ε, σχέση, την αντίληψη για τη σχέση μεταξύ Αρμενίων και Τούρκων. Κατά την άποψή μου το σημείο αυτό είναι ισχυρό σημείο. Νομίζω ότι ε, πλήττεται από τη μνήα στην ε, αρμενική γενοκτονία. Η αναφορά γεγονότων του παρελθόντος δεν η μία αναφορά της ε, γενοκτονίας ε, στην ουσία είναι εις βάρος και της ιστορικής πραγματικότητας και των δικών μας προγενέστερων θέσεων. Ένα άλλο, αν θέλουμε να περάσουμε ένα σαφές μήνυμα για τις μεταρρυθμίσεις, για την συνέχιση του εξυγχρονισμού, θα έπρεπε ωστόσο να ξαναπούμε στους Τούρκους και, σε και κάποιοι διανοούμενοι από την Τουρκία το καταλαβαίνουν, ότι θα πρέπει να μπορούν να ξεπεράσουν και την ιστορία τους και να αναγνωρίσουν το παρελθόν τους. Θα ήθελα να συμπεριληφθεί το σημείο αυτό σε όλη την έκθεση. Ευχαριστώ. Merci. Mr. Ο κύριος Καζάκα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Και εγώ από πλευρά μου θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για την έκθεση που η κυρία Ομενόιτεν και τον ισορροπημένο τόνο που διατηρεί στο κείμενο. Ξέρουμε ότι το θέμα αυτό για τις σχέσεις με την Τουρκία είναι ένα θέμα πολύ ευαίσθητο για πολλούς συναδέλφους. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι η έκθεση έρχεται σε μια πολύ σημαντική στιγμή. Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου πρέπει να πούμε εκ νέου σαφώς αυτό που περιμένουμε από την Τουρκία, ούτω ώστε να πληρεί τα κριτήρια προσχώρησης της Κοπενχάγης. Ωστόσο θέλω να κάνω κάποιες παρατηρήσεις για τις συμβαστικές προτάσεις που θα πρέπει να προταθούν. Σε ό,τι αφορά την συμβιβαστική τροπολογία 2, ε, είμαι πλήρως ικανοποιημένος από την διατήρηση της πρόσκλησης προς την τουρκική πλευρά να εγκριθεί εν τέλει η νομοθεσία για τον διαμεσολαβητή. Είναι ένα σημαντικός, πολύ σημαντικός νόμος για την προστασία των δικαιωμάτων των Τούρκων πολιτών και είναι μια αναγκαιότητα που καθίσταται όλο ένα και πιο επίγουσα στην Τουρκία. Συμβιβαστική τροπολογία 3. Νομίζω ότι υπάρχει μια σύγχυση ε, ε, κακό ε, αναφερόμενη στην περίπτωση της Λεϊλά Ζανά σε ό,τι αφορά τον τομέα της ελευθερίας έκφρασης. Όλοι γνωρίζουμε ότι η Λεϊλά Ζάνα διώκεται όχι για τις ε, απόψεις της με βάση το άρθρο 301 του ποινικού κώδικα αλλά με βάση το άρθρο 314 για, για τρομοκρατικές ε, δραστηριότητες για δραστηριότητες δηλαδή υποστήριξης του ΠΚΚ. Εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε λάβει σαφή θέση κατά του ΠΚΚ ως τρομοκρατικής οργάνωσης. Γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μια διάκριση στο θέμα αυτό. Θα ήθελα επίσης να ασχοληθώ με το θέμα της Κύπρου. Πιστεύω ότι το θέμα της Κύπρου είναι πολύ σημαντικό ζήτημα θα πρέπει να καλέσουμε τις δύο πλευρές να συνεχίσουν καλόπιστα τις διαπραγματεύσεις ελπίζοντας να φτάσουν γρήγορα σε ένα θετικό και για τις δύο πλευρές αποτέλεσμα. Νομίζω ωστόσο ότι πρέπει να καλέσουμε όχι μόνο απόσυρση για απόσυρση των τουρκικών δυνάμεων αλλά και όλων των άλλων δυνάμεων που βρίσκονται επί τόπου. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ελληνικές δυνάμεις και βρετανικές στρατιωτικές δυνάμεις εκεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιτρέψουμε και στις δύο πλευρές να ε, κάνουν παραχωρήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γεωργίου. Ο κύριος Γεωργίου, δύο λεπτά. Ναι, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν να συγχαρώ την κυρία Όμεν. Η έκθεση αποτελεί Μικρόφωνο σα, δεν ακούγεται κύριε Γεωργίου. Έχω τον λόγο τώρα. Λέγω, ε, να συγχαρούμε τώρα την κυρία Όμε. Πράγματι, η έκθεση αποτελεί επιτυχημένη άσκηση ισορροπίας. Θα αναφερθώ σε δύο ε, σημεία. Πρώτον, στο κάζους Μπέλη. Πρέπει να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι αυτό αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία. Εγώ δηλαδή, με 40 χρόνια διπλωματίας πίσω μου, τέτοιο, τέτοιου είδους απειλή δεν την έχω ξανασυναντήσει. Δηλαδή δεν την έχω συναντήσει έστω και σε ταπεινότερες πολιτικές πρακτικές. Έχουμε παραδείγματα όπου οι σχέσεις κρατών έχουν φτάσει στο χείλος του πολέμου και εν τούτης απεφεύγεται αυτή η απειλή εναντίον κράτους το οποίο μάλιστα υποστηρίζει την ένταξη της Τουρκίας στον Ευρωπαϊκό Κορμό. Αυτού του είδους οι απειλές δεν ακούγονται ούτε σε κύκλους του υποκόσμου. Πώς να δεχθώ ότι εκτοξεύονται από ένα οποιοδήποτε σοβαρό κράτος με ευρωπαϊκές προοπτικές. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Το δεύτερο ζήτημα είναι το ζήτημα του χρόνου. Είχατε μιλήσει, ε, ε, ε, είχατε αποφασίσει για το 2009. Αυτό θα υπήρχε καταληκτική ημερομηνία. Να προσέξετε διότι εάν σήμερα εφαρμόσετε άλλου είδους τακτική αυτό θα αποτελέσει υποθήκη και να ξέρετε ότι θα το συναντήσετε ε, μπροστά σας και σε επόμενες ενδεχομένως αιτήσει κρατών που θα ζητήσουν παρόμοιες παρατάσεις. Σε ό,τι αφορά τώρα το ζήτημα της Κύπρου πρέπει να σας πω ότι και αυτό αποτελεί μια άλλη πρωτοτυπία. Εδώ έχουμε δύο προέδρους οι οποίοι πασχίζουν να βρουν μια λύση περί των Κυπριακών και εσείς και εδώ ακούγεται στην αίθουσα που είναι επιτέλους και το πολυτελέστερο φροντιστήριο, φροντιστήριο πολιτικής αυτής της Υπήρου ακούμε κουβέντες για, κόφια, για, για, για ε, ε, σχέδιο Ανάν που τα βρήκατε, που τα ε, βγάλατε αυτά όταν επιτέλους έχουν δοθεί απαντήσεις δια δημοψηφισμάτων αυτά επιτέλους πρέπει να γίνουν μαθήματα όταν κάποιοι αποφασίζουν κάτι νομίζω ότι αυτό πρέπει να τηρείται και να εκτιμάται δεν μας άρεσε το αποτέλεσμα time, του, του, σχεδίου Ανάν το απορρίπτουμε Ευχαριστώ κύριο Ζαλέσκη για μισή λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα αγγλικά. Ριάν, ήθελα να σου κάνω κομπλιμέντο. Θα σου έλεγα ότι με το κείμενό σου, με το περιεχόμενο, με τον τρόπο που το συνέταξες έκανες πολύ μεγαλύτερη πρόοδο από ότι η Τουρκία. Λοιπόν, θα συνεχίσω στη γλώσσα μου. Λοιπόν, όσον αφορά αυτά που έλεγε ο κύριος Σιμάνσκι και αυτό από τη δική μου εμπειρία στο Κοινοβούλιο όσον αφορά την ψηφοφορία για την έκθεση Μπροκ. Πρέπει να πω ότι ελπίζω ότι δεν θα κηρύσουμε στην Τουρκία ότι πρέπει να γίνει κοσμική χώρα, να είναι κοσμική χώρα. Θέλουμε η κυβέρνηση να είναι κοσμική και να ακολουθεί την κοσμική νομοθεσία. Οι τροπολογίες 24, 26, 28 και 31 κάνουν ένα τέτοιο κήρυγμα Κυρίως οι σοσιαλιστές περιμένουν και ελπίζουν ότι πρόκειται να είναι κοσμική χώρα η Τουρκία. Δεν έχουμε το δικαίωμα να ζητούμε κάτι τέτοιο από μια χώρα. Είναι κυρίαρχη χώρα και η χώρα αποφασίζει μόνη της. Εγώ ε, δεν το λέω υποστηρίζοντα το Ισλάμ ή όντας κατά του Ισλάμ. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τη θρησκεία μιας χώρας και για να έχουμε καλύτερη ισορροπία η τροπολογια 64 64-65 είναι πάρα πολύ ήπιες. Εκφράζουμε τη λύπη μας διότι η Τουρκία δεν είναι ανεκτική όσον αφορά τις άλλες θρησκείες. Εγώ θα απαιτούσα να υπάρχει ισοτιμία και ανοχή. Πρέπει να απαιτούμε η χώρα να αντιμετωπίζει έτσι τις άλλες θρησκείες. Σχεδόν τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Πρέπει να είναι ισορροπημένο το κείμενο. Δεν θα πρέπει να κηρύσουμε τι μορφή πρέπει να έχει η χώρα, αν θα είναι κοσμική ή όχι. Πρέπει να αποφασίσει από μόνη η Τουρκία. Αυτά και ευχαριστώ. Η ε, κυρία Ποσκουίτ, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω να πω ένα-δύο πράγματα, λέει η κυρία Μποσκούρτ. Καταρχάς να ευχαριστήσω την κυρία Όμεν Ράιτεν που έλεβε υπόψη αρκετά σημαντικά σημεία όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών μεταξύ άλλων στις τροπολογίες και που υποστήριξε και κάποιες άλλες τροπολογίες που υπευλήθησαν. Ένα πολύ σημαντικό σημείο αφορούσε τις μεταρρυθμίσεις στην Τουρκία. Δηλαδή ότι η Συνταγματική Επιτροπή στην Τουρκία αποφάσισε να δημιουργήσει μια επιτροπή ίσων ευκαιριών στο τουρκικό κοινοβούλιο. Η απόφαση αυτή αναμένεται να ληφθεί σήμερα. Ελπίζω να μπορεί να συμπεριληφθεί αυτό το στοιχείο στην έκθεση. Πέραν αυτού, όσον αφορά της συνεργασία στο δικαστικό τομέα. Συνεργασία μεταξύ δικαστηρίων είναι κάτι πολύ σημαντικό, κυρίως όσον αφορά κάποια ε, Ισλαμικά ιδρύματα και τις γυναίκες. Καμιά φορά ε, οι γυναίκες είναι θύματα. Χρειάζεται καλή συνεργασία μεταξύ τουρκικών αρχών και ευρωπαϊκών αρχών στη δικαστική συνεργασία ώστε να προστατεύουν τα δικαιώματα των ανθρώπων και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Τουρκία και θα πρέπει αυτό να το προσέχουμε όλος ιδιαίτερος και να επιμείνουμε επιβελτιώσεων. Τέλος, θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να προσέξουμε όλος ιδιαίτερος το άρθρο 13 της Ευρωπαϊκής Συνθήκης για τη μη διακριτική μεταχείριση να μην υπάρχει διάκριση για κανένα λόγο αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όσον αφορά την απειλή να κλείσουν κάποια ιδρύματα στην Τουρκία και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα πρέπει η Τουρκία να αποφύγει η αδίποτε διάκριση είτε βάση εθνοτικής καταγωγής γλώσσας, θρησκείας, σεξουαλικής προτίμησης κλπ. Έχω έξι αγορητές, ο καθένας από ένα λεπτό. Ο κύριος Κυρίτα έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, να ευχαριστήσω την κυρία ο Μενερόιτε για την πάρα πολύ καλή εκθεσή της. Καταρχάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ενθαρρύνει την Τουρκία να συνεχίσει την προευρωπαϊκή πορεία της, ε, η οποία θα είναι κοσμική και θα πρέπει να κάνει ε, μεταρρυθμίσεις ποιοτικές ε, προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης θα πρέπει να διασφαλίσει την αυτονομία των πανεπιστημίων και να προσπαθήσει να εντάξει τους φοιτητές της στα προγράμματα Εράσμους. Θα πρέπει επίσης να τους ενθαρρύνουμε να προχωρήσουν τα διάφορα προγράμματα που έχουν. Όσον αφορά τώρα τα δικαιώματα των ανθρώπων και των μειονοτήτων, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να καταδικάσει οποιασδήποτε διαχωριστικές ε, και εθνικιστικές δράσεις. Τα όσα συμβαίνουν στην Τουρκία ε, με το θέμα της Κύπρου είναι ένα παράδειγμα. Θα πρέπει να τηρούνται οι αρχές ε, της εδαφικής κυριότητας και η Τουρκία θα πρέπει ε, να λύσει το θέμα στην περιοχή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κοπάκη, για ένα λεπτό. αρχικά την κυρία Ουμερόιτεν για μια εξαιρετική έκθεση, ουσιαστική και ισορροπημένη. Στηρίζουμε την ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας, πιστεύοντας ότι μόνο αυτή η προοπτική τη βοηθάει στην πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και στη διατήρηση σχέσεων καλή γειτονίας. Αξίζει πιστεύω να παρακολουθήσουμε στενά τις εξελίξεις στην υπόθεση Εργένικων και ελπίζω η τουρκική δικαιοσύνη να φτάσει την υπόθεση στην άκρη γιατί η πλήρης διαλεύκανση είναι μεγάλη πρόκληση για τη χώρα. Η Τουρκία βρίσκεται σε μια κρίσιμη μεταβατική περίοδο τόσο εσωτερικά όσο και σε σχέση με τον επαναπροσδιορισμό του γεωστρατηγικού της ρόλου στον Κάφκοσο και τη Μέση Ανατολή. Και η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να στηρίξει μια Τουρκία η οποία θα μπορεί να λειτουργεί σταθεροποιητικά. Δεν μπορώ όμως να μην επισημάνω ότι οι τελευταίες στρατιωτικές κινήσεις της Τουρκίας στο Αιγαίο δεν διευκολύνουν το διάλογο και δημιουργούν ένα νέο κλίμα έντασης με την Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς πιστεύω ότι η αναφορά της εισηγήτριας στην ανάγκη άρσης του κάζου Ζουσμπέλη μέσα στην τουρκική εθνοσυνέλευση είναι πάρα πολύ σημαντική και πρέπει να διατηρηθεί. Ανταποκρινόμενη στην παράκληση της ηγήτριας για να μην διαταραχθεί η έκθεση, αποσύρω τι τροπολογίε μου 3, 4, 10 και 51. Διατηρώ την τροπολογία 99 για την προστασία των δικαιωμάτων σημερινών και παλαιών μειονοτήτων, καθώς και την 162 που εκφράζει την ανησυχία για την απόφαση κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στο Ακούγιο, που είναι μια σεισμογενής περιοχή. Τελειώνοντας, σχετικά με την Κύπρο, θέλω να τονίσω ότι η λύση με παρουσία στρατευμάτων κατοχής είναι μια πολύ δύσκολη λύση. Ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, κύριος Κασουλίδης, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Δεν θα είχα ζητήσει το λόγο, γιατί η κυρία Ρία Όμεν έχει διαχειριστεί το ζήτημα με πάρα πολύ καλό τρόπο. Θα ήθελα να πω δύο διευκρινιστικά πράγματα σε δύο συναδέλφους. Ε, πρώτον, το, προς τον κύριο Λάκεντάικ. Το θέμα των θεμελιωδών ελευθερών όσον αφορά τις προσωρινές παρεκκλήσεις είναι κάτι το οποίο δέχεται το ευρωπαϊκό κεκτημένο και οι αρχές βάσει των οποίων θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι οι μόνιμες παρεκκλήσεις από τις βασικές ελευθερίες. Και φρονώ ότι όταν ε, κάνουμε διαπραγματεύσει ε, στην Κύπρο, έχουμε κατά νου τι προσωρινέ παρεκκλήσει. Εμεί είμαστε οι πρώτοι που θέλουμε λύση του προβλήματό μα και δεν θα είχαμε ποτέ εισαγάγει κάτι το οποίο θα παρακόλλει τη λύση. Ω προς το όσα είπε ο κύριο Βόμποντα, δέχομαι του φόβου ε, τη διαδικασία ε, όσον αφορά την ημερομηνία του Δεκεμβρίου του 2009. Και για να μην έχουμε περαιτέρω ε, συνέπειες για τις διαπραγματεύσεις θα μπορούσαμε ίσως να χρησιμοποιήσουμε τον όρο may ε, για να μην έχουμε περισσότερα προβλήματα. Δεν ξέρω αν συ, συμφωνεί ο κύριος ε, Σβόμποντα. Ευχαριστώ πολύ λέει κυρία κυρία Μπεγκέν. Ε, εδώ βλέπω να περιορίζεται όλο και περισσότερο χρόνο. Θα ήθελα να σταθώ στο θέμα της ε, πολιτικής γειτονίας και να συγχαρώ και την κυρία Ομεν Ρόιτεν για την εργασία της. Η Τουρκία διαδραματίζει ένα πάρα πολύ σημαντικό ρόλο αυτή τη στιγμή σε ό,τι αφορά τη διαμετακόμιση ενέργειας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης για την εξασφάλιση της σταθερότητας της περιοχής του Νότιου Καυκάσου. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια και να της θέσω το ερώτημα του κατά πόσο θα μπορούσε να ενσωματώσει και τις προτάσεις που έχουν γίνει από την ομάδα μας σε σχέση με τον ρόλο που έχει διαδραματίσει η Τουρκία στα πλαίσια της σύγκρουσης της Γεωργίας και της Ρωσίας προσπαθώντας να επιτύχει τη συμφιλίωση των δύο πλευρών και επίσης θέλω να τονίσω αυτό το κομμάτι της εκθέσεως αλλά δεν έχει τονιστεί ή εξηγηθεί επαρκώς ότι εμείς θα πρέπει να επιμείνουμε η Τουρκία να ανοίξει τα σύνορά της με την Αρμενία, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο ζητούμε από την αρχή. Δεν είναι μια, ένα προαπαιτούμενο μεν, αλλά δεν μπορούμε να φανταστούμε μια χώρα η οποία βρίσκεται σε στάδιο προενταξιακό και εξακολουθεί να κρατάει κλειστά τα σύνορά της με τις όμορες χώρες. Κάτι τέτοιο λοιπόν θα επέτρεπε και την χαλάρωση των εντάσεων και να βρεθεί και κάποια συμβαστική λύση μεταξύ Αζερμπαϊτζάν και Αρμενίας για το Άνω Καραμπάχ. Ο κύριο Τάνοκ, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θέλω να συγχαρώ τη Ρία Όμεν και Ρόιτεν για τη θαυμασία έκθεσή τη. Δεν θα μιλούσα, αλλά έχω κάποια αντίρρηση για τα σχόλια του κυρίου Καζάκ σε σχέση με τα 45.000 στρατεύματα της ε, Τουρκίας στη Βόρεια Κύπρο και την παρουσία Βρετανικών στρατευμάτων στην Κύπρο, στη Δημοκρατία της Κύπρου. Δεν υπάρχει ούτε ένας φαντάρος στην Κύπρο. Είναι στην κυρίαρχη βάση Στι κυρίαρχε βάσει, όπω προβλέπεται από τι συνθήκε του 1960. Είναι εκτό του εδάφους Κυπριακή Δημοκρατία, Δημοκρατίας, εκτός Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι μόνοι στρατιώτε στη Δημοκρατία Κύπρου είναι αυτοί που βρισκόνται στην ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ. Υπάρχει μια μικρή ελληνική δύναμη χιλίων στρατιωτών βάσει τι ε, του 1960 και 650 Τούρκοι στρατιώτε, Εκεί θα πρέπει να ξαναγυρίσουμε και όχι στους 40.000 οι οποίοι είναι η δύναμη κατοχή στο βορρά. Η Τουρκία δεν φαίνεται ποτέ να βρει την ευκαιρία να κάνει σωστές δημόσιες σχέσεις. Παραδείγματος χάρη γιατί δεν έχουν ακόμα ανοίξει την ε, σχολή της Χάλκης, την ελληνοορθόδοξη σχολή, παρά τις επανειλημμένες αιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που έπεσαν σε κοφά ότα. Και θα ήθελα να επενθυμίσω στην κυρία Σλερμπεκέν την παράγραφο 57 για τα απογοητευτικά αποτελέσματα από την επίσκεψη του Προέδρου Γκιουλ στην Αρμενία. Δεν υπήρξε καμία πρόθεση στι διμερεις σχεσει σκέψεις, σχέσεις Αρμενίας-Τουρκίας. Είναι ακόμα παγωμένε οι σχέσει, πρέπει να περνάνε από τη Γεωργία οι εμπορικέ ροέ. Επομένω, θέλω να τονίσω και πάλι ότι η Τουρκία πρέπει να δείξει καλή θέληση με το να ανοίξει τα σύνορά τη με την Αρμενία. Πριν δώσω τον λόγο στην εισηγήτρια, θα ζητήσω από τον κύριο Φιλόρη να κάνει κάποιο σχόλιο από τη Γενική Διεύθυνση διεύθυνση. Button on the right Το, το κουμπί στα δεξιά σας. Excuse Συγγνώμη. Η Επιτροπή θέλει να ευχαριστήσει ιδίως και θερμά την κυρία Όμεν για την εξαιρετική και σημαντική δουλειά που έκανε με την έκθεση. Όπως πάντα, κυρία εισηγήτρια, η έκθεση είναι πλήρης, λεπτομέρειας που αντικατοπτρίζει τα ευρήματα της έκθεσης επιτροπή για το 2008. Με τρει παρατηρήσει, παρατηρήσεις σύντομες θα κάνω μετά την συζήτηση που ακούσαμε. Πρώτον, υπάρχει από ό,τι φαίνεται και το διαπιστώνουμε και εμείς νέο κλίμα στην Τουρκία ή τουλάχιστον μια νέα προσπάθεια νέα εκκίνηση των, μετα... των μεταρρυθμιστικών σπαθιών μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Ερντογάν στις Βρυξέλλες και την επίσκεψη του αρχηγού τη αντιπολίτευσης χτες υπάρχει σαφή δέσμευση από πλευράς Τουρκίας να τηρήσει τον δρόμο των μεταρρυθμίσεων εν ώψη της προσχώρησης. Κατά την άποψή μας θα έπρεπε το κλίμα αυτό να αντικατοπτρίζεται και στην έκθεση. Δεύτερο θέμα η καταληκτική ημερομηνία του Δεκεμβρίου του 2009. Υπενθυμίζω ότι το, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2006 έλεγαν ότι η Επιτροπή θα αναφέρει σε, για όλα τα, σημαντικά ζητήματα για το 2007, 2008 και 2009. Το ίδιο το Συμβούλιο δεν προδίκασε την έκβαση των συζητήσεων που θα λάβουν χώρα στο τέλος του έτους. Η συζήτηση αυτή θα γίνει εν ευθέτω χρόνο, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ε, σημαντικά συναφή στοιχεία. Και είναι σημαντικό να μην προδικάζουμε με οποιοδήποτε τρόπο την έκβασή τους. Εμείς στην Επιτροπή δεν κάνουμε καμία δημόσια δήλωση σχετικά προσπαθώντας να αποφύγουμε το να προδικάσουμε τις σχετικές συζητήσεις. Δεύτερο θέμα, Κύπρος. Θέλω να αναφέρω, να παραθέσω, δεν θα σχολιάσω το σχέδιο Ανάν που απορρίφθηκε όντως, αλλά θα αναφερθώ στο 10ο πρωτόκολλο της πράξης προσχώρησης του 2003. Το 10ο πρωτόκολλο λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να ε, αντιμετωπίσει την ε, συνολική λύση του Κυπριακού με βάση τις γραμμές πάνω στις οποίες ε, θεμελιώνεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μιλώντας κυρίως για το άρθρο 6 της συνθήκης που αφορά την τήρηση του κράτους δικαίου, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της δημοκρατίας. Και εδώ, ως Επιτροπή, απέχουμε από οποιαδήποτε κρίση που θα προδίκαζε την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο νησί για όλες τις άλλες πτυχές που θα αντιμετωπιστούν κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Και δεν συμπεριλαμβάνουμε, κατά την άποψή μας, μεταξύ των θεμελιωδών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέματα που αφορούν στις τέσσερις ελευθερίες. Κάτι σημαντικό για να επιτρέψουμε στους διαπραγματευτές των νησί να έχουν αρκετό περιθώριο συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Είναι ένα θέμα που θα διευκρινίσουμε βάσει του πρωτογενούς δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά βάση της συνθήκης προσχώρησης του 2004. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Φιλόρη για την άποψη Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Άμεν Ράιτεν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ για όλες τις παρατηρήσεις που έκαναν οι συνάδελφοί μου. Καταρχάς ε, θα ήθελα να απαντήσω γενικά. Πρώτα απ' όλα νομίζω όσον αφορά την τροπολογία 36 Ιωάννης Βόμποντα θα μπορούσαμε να κάνουμε προφορική τροπολογία. Θα μπορούσαμε να έχουμε ένα νέο κείμενο που θα προτείνω για την ψηφοφορία σήμερα το απόγευμα. Όσον αφορά την προθεσμία του 2009, νομίζω ότι ο κ. Κασουλίδης με τα σχόλιά του αναφέρθηκε στο θέμα. Παίρνω το κείμενο όπως θα μπορούσε να διατυπωθεί. Στην παράγραφό μου 27 και απαντώ και στον κύριο Φιλόρη λέγοντας αυτό, υπενθυμίζει ότι μία εκπλήρωση των δεσμεύσεων της Τουρκίας μέχρι τον Δεκέμβριο του 2009 ίσως σοβαρά να επηρεάσει τις διαπραγματευτικές διαδικασίες. Θα μπορούσα πραγματικά να δεχτώ ένα τέτοιο κείμενο και για μία ακόμη φορά θα ήθελα να τονίσω απευθυνόμαστε στον κύριο Φιλόρη ότι σε αυτό το κείμενο δεν υπάρχει καμία προκατάληψη, δεν προδικάζουμε κάτι. Απλώς επαναλαμβάνω τα όσα ήδη έχει πει και έχει κάνει το Συμβούλιο. Χαίρομαι που και οι σοσιαλιστές μάλλον μπορούν να το δεχτούν αυτό. Ευχαριστώ τα, τους φιλελευθέρους για τα σχόλια τους όσον αφορά την απόσυρση των στρατευμάτων από την Κύπρο και το σχετικό κείμενο. Δεν θέλω να το αλλάξω αυτό το κείμενο. Γιατί? Διότι αν το αλλάξω πολλοί άλλοι συνάδελφοι θα έχουν ε, νέα προβλήματα. Σε αυτό το κείμενο, ε, αν το διαβάσετε πολύ προσεκτικά, καλό την Τουρκία να διευκολύνει τη δημιουργία κλίματος για διαπραγματεύσεις αποσύροντας τουρκικές δυνάμεις. Ε, δεν ζητώ να αποσυρθούν όλα τα τουρκικά στρατεύματα. Δεν ζητώ κάτι τέτοιο. Ελπίζω και να αφήσουμε τους δύο ηγέτες να πραγματοτευθούν ελεύθερα για το μέλλον των χωρών τους. Είναι πιο ανοιχτό το κείμενο από αυτό που πιστεύει ο κύριος Λάγκεντάικ. Ο κύριος Σιμάνσκι, ναι, στη συμβαστική τροπολογία 5 αναφέρομαι και στις αρχές των συνθήκών μας. Ελπίζω να κανοποίησα τον κύριο Λάγκεντάικ όσον αφορά τις διευθετήσεις για το ελεύθερο εμπόριο. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να φέρουμε ε, στην τράπεζα των υπαγματεύσεων στην Τουρκία και να διαπραγματευτούμε όπως διαπραγματευόμαστε τρεις τρίτες χώρες. Μπορούν να γίνονται παράλληλες διαπραγματεύσεις, αλλά δεν είναι ακόμα μέλος της ενώσεως δεν μπορεί να είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Αυτό είναι ανέφικτο. Ελπίζω να εξηγώ αυτή την τροπολογία. Έχουμε αρκετές τροπολογίες και ΕΓΕ. Γιατί ζήτησα να καταψηφιστούν κάποιες τροπολογίες σας. Πρώτα απ' όλα, επαναλαμβάνετε τα ήδη υποθέντα. Αυτά που αναφέρονται στην έκθεση και δεν θέλω να ψηφίσουμε χριστουγεννιάτικο δέντρο. Γι' αυτό καταψηφίζω κάποιες από τις τροπολογίες σας. Υπάρχουν όμως και τροπολογίες που ε, είναι αδικαιολόγητες θα έλεγα, τεκμηρίωτες, όπως η 116 για τις ποσοστώσεις για τις μεταφορές. Αυτό δεν είναι θέμα ευρωπαϊκό αλλά διμερές. Γι' αυτό πρέπει να καταψηφίσω την εν λόγω τροπολογία και σας παρακαλώ να έχετε υπόψη σας ότι όλα όσα έκανα έχουν ελεγχθεί. Έχουν ελεγχθεί. Λοιπόν, Πρόεδρε, ελπίζω ότι ο κ. θα αποσύρει αυτές τις τροπολογίες που ζήτησαν να αποσύρει. Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι έθεσαν ερωτήσει, χρειάζεται να απαντήσω άλλους, σε άλλους, γιατί πρέπει να προχωρήσω γρήγορα. Μάλιστα. Ο Τσάρλ Τάνοκ και άλλοι που έκαναν σχόλια σχετικά με την παράγραφο περί Αρμενίας. Τι κάνω. Προσθέτω, προσθέτω κάποια σημεία στις παραγράφους που ήδη ψηφίσαμε τις περασμένες δύο-τρεις φορές. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν καλές σχέσεις μεταξύ Αρμενίας και Τουρκίας. Επίσης πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν είναι πρόεδρος Γκιούλ που επισκέφθη την Αρμενία, αλλά γίνονται και άλλα βήματα έγιναν του τελευταίους μήνες και άλλα βήματα που δημιουργούν ελπίδες για μας ότι θα εξομαλυνθούν οι σχέσεις. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι σας παρακαλώ μην πειράζετε αυτή την προσεκτικά διατυπωμένη παράγραφο διότι δεν έχει νόημα κάτι τέτοιο. Αυτά και ευχαριστώ Πρόεδρε. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Θα ψηφίσουμε σήμερα το απόγευμα στις 4.30.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

Uh, Παρακαλώ. όλους, εάν θέλουν να φύγουν, να φύγουν ησύχως και ηρέμος. Dear colleagues, uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, yeah. προχωρούμε στο σημείο υπαριθμό 14 της μέσης διαταξής μας. Είναι η αντιλαγή απόψε με τον κύριο Φέιθ, ο οποίο είναι ο ειδικό μας εκπρόσωπος στο Κωσυφοπέδιο. Τον καλωσορίζουμε και φυσικά δεν είναι η πρώτη φορά. Το Κωσυφοπέδιο είναι κομβική σημασία σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρία Φέιθ η παρουσία σας εδώ σηματοδοτεί δύο σημαντικά ορόσημα. Το γεγονός ότι σας ε, διορίσανε τον Φεβρουάριο του 2008 στο αξίωμά και επίσης τα γενέθλιά σας που νομίζω ότι ήταν την περασμένη Δευτέρα, όπως με πληροφόρουν. Και σας εύχομαι χρόνια πολλά. Φαίνεται λοιπόν ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στο κοσφοπέδιο είναι μεγάλες και πολλαπλές αλλά είστε ακόμα νέος και δραστήριος. Είναι δραστηριότητες μεγάλης εμβέλειας. Η εκπροσώπηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από εμάς στο Κωσυφοπαίδιο έχει σαν στόχο να εξασφαλίσει ότι η αποστολή EULEX που είναι η μεγαλύτερη αποστολή στα πλαίσια της ΚΕΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης λειτουργεί σωστά, ότι διατηρείται το κύρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης εναντί όλων των συνομιλητών μας και ότι φυσικά θα εκπληρωθεί η τριπλή εντολή να προωθήσετε τη δημιουργία μιας αποτελεσματικής, ανεξάρτητης, πολυεθνικής δομής στο κοσμοπεδίο Δεύτερον, να αντιμετωπίσετε το οργανωμένο έγκλημα <clears throat> και τη διαφθορά. Και τρίτον, <clears throat> να αντιμετωπίσετε το άχθος του παρελθόντος το οποίο εξακολουθεί να σκιάζει αυτό το τμήμα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να φέρετε τους υπευθύνους ενώπιον της δικαιοσύνης για τα εγκλήματα του παρελθόντος. Πρέπει επίσης να συνεργαστείτε με τις αρχές του κοσμοπεδίου για να εξασφαλίσετε ότι πράγματι θα εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Σύνταγμα, ιδίως σε ό,τι αφορά την προστασία των μειονότητων και ιδίως της σερβικής μειονότητας και ξέρετε ότι μπορείτε να βασίζεστε στην πλήρη υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχόμεθα κάθε επιτυχία στο έργο σας. Έχουμε εγκρίνει την προηγούμενη εβδομάδα ένα ψήφισμα <clears throat> που δίνει την πλήρη υποστήριξή μας στο έργο σας και σας ενθαρρύνει να συνεχίσετε τις προσπάθειές σας. Κύριε Φέη, θα ήθελα λοιπόν να έχουμε την αξιολόγηση του έργου σας μετά από τον πρώτο χρόνο παρουσία σας και την αποτίμηση αυτών που έχει πράξει μέχρι τώρα κυβέρνηση του Κωσυφοπέδιου και των προκλήσεων που παραμένουν ενώπιόν μας και επίσης να μας πείτε ποια είναι και η επιτόπια κατάσταση, ιδίω πώς λειτουργεί και αναπτύσσεται η αποστολή της ULEX και αν έχει περατωθεί, αν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξή της και επίσης η αντιμετώπιση του προβλήματος των θυλάκων των Σέρβων και στο βορρά και στο νότο και να μας πείτε πώς υπάρχει συνεργασία από το, από το Βελιγράδι για την αποστολή της ε, Ulex αν διευκολύνει τη λειτουργία της Ulex και τα συναφή θέματα. Έχετε το λόγο κύριε Φέιθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια. Για μένα προσωπικά. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρίες και κύριοι, Χαίρο που είμαι εδώ μαζί σας σήμερα για να σας παράσχω την εκτίμησή μου για την πρόοδο που επιτεύχθηκε, για την στερέωση και το συντονισμό της ευρωπαϊκής παρουσίας στο κοσφοπέδιο, καθώς και για τις πρωτοβουλίες που ανέλαβα ως τμήμα των εντεταλμένων ευθυνών μου σχετικά. Είναι και επίκαιρη η στιγμή που έρχομαι εδώ, όχι μόνο λόγω των γενεθλίων που αναφέρατε, αλλά και διότι έρχεται, πιο σημαντικό, από την έγκριση, μετά την έγκριση στις 5 Φεβρουαρίου από το Κοινοβουλίο, ενός ψηφίσματος για το κοσυφοπαίδιο και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διάβασα το ψήφισμα όπου αναφέρεται το Κοινοβούλιο εκφράζει την πλήρη υποστήριξή της στην αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κοσφοπέδιο στις προσπάθειες της αποστολής να συνεργαστούν με τις αρχές στην Πρίστινα για την ευρωπαϊκή προοπτική του Κοσφοπέδιου ως τμήματος της περιοχής. Ενώ αναφέρει επίσης ότι πρέπει να υπενθυμίζουμε στις αρχές της Πρίστινα τις δεσμεύσεις της ιδιαίτερα για την ενίσχυση του κράτους δικαίου και την συνέχιση του σεβασμού του σεβασμού των κοινοτικών δραστηριοτήτων. Καλωσορίζω ιδιαίτερα την υποστήριξη που δίδει το ψήφισμα από αυτό σε μένα για βασικά θέματα όπως την αποκέντρωση, την προστασία της θρησκευτική και πολιτισμικής κληρονομιάς, την οικονομική μεταρρύθμιση και τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της ασφάλειας. Θα επανέλθω στα θέματα αυτά με περισσότερες λεπτομέρειες αργότερα στην παρουσίασή μου. Η υποστήριξή σας σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς δουλειάς ε, μου δίνει τη δυνατότητα για να παλέψω ακόμα σκληρότερα για να υπάρξει γρήγορη πρόοδος και φέτος και πέραν του 2009. Στην παράγραφο 32 του ψηφίσματος πρόεδρε διαπιστώνω ότι το, κείμενο, το Κοινοβούλιο εκφράζει την ανησυχία του για την αργή πορεία των μεταρρυθμίσεων ε, που έχουν ξεκινήσει οι αρχές του κοσφοπεδίου. Όντως, η κυβέρνηση πρέπει να αναλάβει ουσιαστικά βήματα στους τομείς της λογοδοσίας και της διαφάνειας, αλλά και στην μάχη κατά της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Επίσης, πρέπει να ενισχύσει τους δεσμούς μεταξύ πολιτικής και ζωής και κοινωνίας των πολιτών και να, και να χρησιμοποιήσει με υπεύθυνο και ανοιχτό τρόπο τα δημόσια και τα διεθνή κονδύλια. Όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρεται είναι βασικά στοιχεία για να υπάρξει ένα περιβάλλον που θα επιτρέψει την περαιτέρω στερέωση των ευρωπαϊκών προσδοκιών του κοσυφοπεδίου και θα βοηθήσει να βελτιωθούν οι οικονομικές και κοινωνικές ε, συνθήκες στην καθημερινότητα των πολιτών. Πέρυσι, Πρόεδρε, το, κοινο, Κοσμοπέδιο θέτησε ένα σύνταγμα, ενέκρινε νέα σημαντικά νομοθετικά κείμενα, ενίσχυσε βασικά υπουργεία, προώθησε την θέσπιση και έναρξη λειτουργία ενός συνταγματικού δικαστηρίου και άλλων βασικών θεσμών ασφάλειας και ανεξαρτησίας και μετατρέπεται σταδιακά σε κομμάτι της διεθνούς κοινότητας. Οι εξελίξεις αυτές πραγματοποιήθηκαν όλες μέσα σε ένα σχετικά ασφαλές περιβάλλον. Το περασμένο Δεκέμβριο η EULEX ξεκίνησε την αποστολή της στο Κωσυφοπαίδιο και αυτό πετέλεσε ένα σημαντικό βήμα προς το εμπρός για την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως πρωταγωνίστριας ε, στο κοσυφοπέδιο. Αυτή η εξέλιξη επέτρεψε την ενίσχυση τριών βασικών τομέων που είναι κέντρο της δουλειά μας και φέτος και στα επόμενα έτη. Σταθερότητας, μεταρρύθμισης και συμφιλίωσης. Θα αναφερθώ στους στρατηγικούς στόχους σταδιακά και θα κλείσω προτείνοντας τον καλύτερο τρόπο για να πετύχουμε κάτι τέτοιο σε συνεργασία με τις αρχές του Κωσοβερίου. Η βιωσιμότητα των όλων των πρωτοβουλειών εξαρτάται κατά βάση από τη συνέχιση της πολιτικής σταθερότητας του κοσμοπέδιου. Όπως είπα, ενώσο παραμένει, ε, ναι μεν παρέμεινε σταθερή η κατάσταση στο Κωσυφοπέδιο πέρυσι και οι πολιτικές αντιδράσεις της Πρίστινας στις συζητήσεις με, υπό την αιγίδα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι πρόσφατες εξελίξεις στην Μητρόβιτσα δείχνουν πόσο τρωτή και εύθραυστη είναι η κατάσταση επιτόπου. Ως ειδικός αντιπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκίνησα έναν τοπικό μηχανισμό ε, ανοιχτών διαβουλεύσεων για θέματα πρακτικής σημασίας, όπως μεταξύ των οποίων θέματα που αναφέρονται και στην έκθεση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ τον Νοέμβριο του 8. Μεταξύ των σημείων των θεμάτων αυτών περιλαμβάνονται ίσπραξη δασμών και ε, διανομή εισοδήματος, η λειτουργία των δικαστηρίων στη Μητρόβιτσα, το εφαρμοστέο δίκαιο και η λειτουργία των σιδηροδρόμων στο βόρειο τμήμα. Έχω την άποψη και είμαι βέβαιος γι' αυτό ότι αν κρατήσουμε τη συζήτηση σε τεχνικό επίπεδο, αν προωθήσουμε ευρωπαϊκές βέλτιστες πρακτικές και ευρωπαϊκά πρότυπα και αν εμπλέξουμε στενά τους τοπικούς, διεθνούς και ευρωπαϊκούς εμπλεκόμενους, θα υπάρξει πρόοδος και αποτελέσματα σε κάποιους τομείς. Αυτό είναι κομμάτι του στενού συντονισμού και της συνεργασίας με τον επικεφαλή της ε, αποστολής της EULEX, τον στρατηγό Δεκαμομπών και κάτι τέτοιο ζητάει και το ψήφισμά σας άλλωστε. Εφόσον η Πρίστινα και το Βελιγράδι ενώνονται σε ένα ευρωπαϊκό μέλλον και η Ευρώπη έχει, αναπέξει, έχει αναλάβει ηγετικό ρόλο, μπορεί εμείς να είμαστε αυτοί που ε, θα λειτουργήσουμε ως γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πρωτευουσών. Αν θέλουμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα, έχουμε επιτόπου τα εργαλεία για να βοηθήσουμε να επέλθει ένα τέτοιο ευκταίο αποτέλεσμα. Ο συνολικός στόχος ωστόσο παραμένει η ύπαρξη απευθείας καλών και φιλικών γειτονικών σχέσεων μεταξύ των δύο πλευρών. Η εμπλοκή στο, με τον τρόπο αυτό θα διευκολύνει και την πλήρη επιχειριακή λειτουργία της Ήγιουλεξ όλο το κοσμοπέδιο το συντομότερο δυνατό. Η απέκτηση αυτή, όπως και η ανάγκη ενίσχυση του κράτους δικαίου, ήταν θέματα που συζήτησαν τακτικά και ο Πρωθυπουργός και αντιπολίτευση και δημόσια και ιδιωτικά σε συναντήσεις όπως και με μένα. Η ανάγκη να προχωρήσουμε γρήγορα, ιδίως στον Βορρά, τονίστηκε ακόμα περισσότερο από τα βία γεγονότα κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων και κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων στην Μητρόβιτσα. Στο πλαίσιο αυτό, κάποια κρίσιμα ε, ζητήματα για την ε, λειτουργία των δικαστικών αρχών και την αντιμετώπιση κάποιων εγκληματιών υψηλού επίπεδου πρέπει να αντιμετωπιστούν. Η απάντηση θα έχει συνέπειες για την αξιοπιστία της Ένωσης και την δυνατότητά της να αναλάβει δύσκολα και επικίνδυνα έργα για να ενσωματώσει τον Βορρά και να εξομαλύνει την κατάσταση εκεί ε, ως τμήματος ενός και μόνο ενιαίου τελωνιακού και δικαστικού χώρου που θα στηρίζεται στις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Οι πολίτες στο Κωσυφοπέδιο προσδοκούν πάρα πολλά πράγματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μπορούμε να τους απογοητεύσουμε και να μην τηρήσουμε τις ευθύνες μας. Σε πολιτικό επίπεδο, και εδώ είναι που τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν να παίξουν ε, κρίσιμο ρόλο, η εντατικοποίηση και η βελτίωση της υποστήριξης στο, του Βελιγραδίου στις επιτόπου ε, ευρωπαϊκές αποστολές έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα ως ό,τι αφορά την ε, ανάγκη να υπάρξει περισσότερη συνεργασία από πλευράς των δημάρχων στο βορρά και ε, η απομόνωση των μεγάλων εγκληματιών στην ίδια περιοχή. Προς την κατεύθυνση αυτή πιστεύω ότι η απόφαση του Προέδρου του Κωσυφοπεδίου να μην διεξαγάγει φέτος πολιτικές εκλογές θα βοηθήσει στην διατήρηση της σταθερότητας στην πολιτική κατάσταση της, της χώρας σε ό,τι αφορά τις δημοτικές εκλογές που θα λάβουν χώρα φέτος δεν έχει ληφθεί μέχρι τώρα τελική απόφαση ως προς το πότε θα πραγματοποιηθούν. Η πρόοδος στην αποκέντρωση και η διασφάλιση της συμμετοχής των Σέρβων θα είναι σημαντικά στοιχεία που θα ληφθούν υπόψη να αποφασίσουμε την ακριβή ημερομηνία. Ένα άλλο μια άλλη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη μιας λειτουργούσας κεντρικής επιτροπής εκλογών. Συνεχίζονται οι σχετικές συζητήσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών. Η κυβέρνηση επιθυμεί να γίνει απογραφή του πληθυσμού σε ολόκληρο το κοσμοπέδιο το συντομότερο δυνατό. Θα μιλήσω, θα συζητήσω με τις αρχές για την ε, χρονική στιγμή. Η πρόσφατη ε, η πρόσφατη απογραφή είχε συμμετοχή 71% των Σέρβων του Κοσμοπεδίου και θέλουμε το ποσοστό συμμετοχή στην απογραφή αυτή να αυξηθεί περαιτέρω. Κύριε Πρόεδρε, η συνέλευση του, του Κοσμοπεδίου έπαιξε βασικό ρόλο στην θεσμική εξέλιξη της χώρας από τη στιγμή που δημιουργήθηκε. Πέραν της υποστήριξης των βασικών θεμελιωδών κειμένων και της κύρωσης του συντάγματος, παίζει βασικό ρόλο στις προσπάθειες των θεσμικών αρχών του Κωσυφοπεδίου να εφαρμόσουν μια σειρά θεσμικών οργανικών νόμων, ιδίω που αφορούν την, ε, τα δικαιώματα των μειονοτήτων. Ωστόσο, συνεχίζω να πιστεύω ότι δεν πληρεί τον βασικό της ρόλο σε μια δημοκρατία η συνέλευση. Να είναι δηλαδή ο κύριος χώρος πολιτικής συζήτησης και κοινοβουλευτικής παρακολούθησης και εποπτείας και ελέγχου. Πολλέ αποφάσεις συνεχίζονται να λαμβάνονται από την κυβέρνηση χωρίς πραγματική εμπλοκή της συνέλευσης. Ε, οι πολιτικές συζητήσεις πολλής, περνούν είτε από τον τύπο είτε από τις διαδηλώσει. Παραμένει νέο όργανο ακόμα και γι' αυτό το λόγο η συνέλευση πρέπει να τύχει πλήρους υποστήριξής μας και μόνιμης υποστήριξής μας. Η απόφαση μη διεξαγωγή των εκλογών ήταν του Προέδρου. Όμως, με σιγουριά μπορώ να πω ότι η αποφυγή των γενικών εκλογών φέτος ε, ε, εξαφανίζει ένα αίτιο απόσπαση προσοχής και μπορεί και το νομοθετικό και οι νομοθετικοί και η κυβέρνηση να κάνουν τις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του στο κοσυφοπαίδιο να σταθεί στα πόδια του και είναι κάτι ζωτικό για μελλοντική πρόοδο να γίνει κάτι τέτοιο. Ξεκινώντας λοιπόν, θα έλεγα ότι η κυβέρνηση υποσχέθηκε την ιδιωτικοποίηση των κρατικών επιχειρήσεων, αλλά ακόμα δεν έχει διατυπώσει μια συγκεκριμένη στρατηγική. Αρχικά σχέδια έχουν ανακοινωθεί σε εμβριακό στάδιο ακόμα για την παραγωγή ε, ηλεκτρικής ενέργειας, για τις τηλεπικοινωνίες και τα ταχυδρομεία, καθώς και για το αεροδρόμιο. Πρέπει να προχωρήσουν αυτά τα σχέδια με καλύτερο ρυθμό, όμως η παρούσα οικονομική ύφεση ίσως ε, μειώσει τις άμεσες επενδύσεις, ξένες επενδύσεις στο κοσυφοπέδιο. Γενικότερα, οι αρχές του κοσυφοπέδιου θα πρέπει να διαχειριστούν τις δημόσιες επιχειρήσεις με διαφάνεια και να διορίσουν τα κατάλληλα άτομα στα διοικητικά συμβούλια βάσει των προσόντων τους και των ικανοτήτων τους και όχι βάσει πολιτικών ε, και κομματικών ε, προτιμήσεων. Στον τομέα της μεταρρύθμισης της, ε, της μεταρρυθμίσεως του τομέα της ασφάλειας τον Ιανουάριο, το 20 Ιανουαρίου άλλαξε η δομή των δυνάμεων ασφαλείας του κοσυφοπεδίου. Αυτή η διαδικασία υπογραμμίζεται και στο ψήφισμά σας και είναι κάτι που επιτρέπει να υπάρχει μια μικρή δύναμη ασφαλείας με καθήκοντα προστασίας των πολιτών και μπορεί επίσης να ε, υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο. Όμως η επιλογή των μελών των δυνάμεων ασφαλείας του Κωσυφοπεδίου πιθανότατα θα δημιουργήσει προβλήματα α, ε, όσον αφορά τα πρώην μέλη του KPC και ίσως να δημιουργηθούν κάποιες εντάσεις εξ αυτού. Και έρχομαι στην τρίτη προτεραιότητα. Υπάρχει ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες για συμφιλίωση μεταξύ των διαφόρων κοινοτήτων του Κωσυφοπεδίου. Όπως μου ζητήσατε να κάνω στο ψήφισμά σας, ενθαρρύνω και υποστηρίζω την ε, ηγεσία του Κωσυφοπεδίου. Θα πρέπει να αυξήσει τις προσπάθειές της για να πλησιάσει τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου και άλλες κοινότητες και ίσως πράγματι τώρα να υπάρχει μια δυνατότητα όλο και περισσότεροι Σέρβοι του Κωσυφεδίου να θέλουν να συνεργαστούν με τους κεντρικούς θεσμούς. Έγινε γύρω σε συζήτηση τρογγυλής τραπέζης πρόσφατα και ξεκίνησε διάλογος επιτυχής για συγκεκριμένα θέματα όπως είναι η υγεία, όπως είναι η παιδεία. Ο Πρωθυπουργό και βασικοί υπουργοί συμμετείχαν και θα παραμείνουν στις συνομιλίες αυτές. Οι ηγέτες των Σέρβων του Κωσουπεδίου και από τον Βορρά εξέφρασαν την προθυμία να υποστηρίξουν αυτή την πρωτοβουλία της οποίας ηγείται ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στον ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της θρησκευτική και πολιτιστικής κληρονομιάς έχει ήδη επιτευχθεί κάποια πρόοδους. Συνεργαστήκαμε στενά με το Υπουργείο Πολιτισμού καθώς και με το γραφείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να βρεθεί ένας τρόπος ανταλλαγής τεχνικών πληροφοριών στους συγκεκριμένους τομείς. Σύμφωνα με την συνεργασία, την Ευρωπαϊκή Τερική Σχέση, θέλουμε να ενισχύσουμε τους μηχανισμούς εκείνους που προστατεύουν την πλούσια θρησκευτική και πολιτιστική κληρονομιά που υπάρχει στο Κωσυφοπέδιο. Η πρώτη συνεδρίαση του Φόρουμ διεξήχθη προ 15 περίπου ημερών και εκεί ήρθαν διάφοροι εκπρόσωποι στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς, η ΟΝΜΙΚ συμμετείχε και το Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλοί άλλοι φορείς και έτσι ε, μπορούμε να κατευθύνουμε σωστά το πολιτικό πρόγραμμα που πρέπει να ακολουθηθεί. Μετά από αυτή την ανακτήρια συνεδρίαση έχει μάλλον δρομολογηθεί μια διαδικασία που θα συνεχιστεί και θα είναι επωφελής για, την, για το κοσυφοπαίδιο και θα ωφεληθεί και από την συμμετοχή ή κάποια υποστήριξη που θα δοθεί από τις ε, σερβικές αρχές και από τη σερβική Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι αρχές επίσης εξακολουθούν να σημειώνουν πρόοδο ε, προετοιμαζόμενες για αποκέντρωση. Πριν από μερικές ημέρες ο Πρωθυπουργό ανακοίνωσε ότι οι αρμοδιότητες για την, για την κοινωνική πρόνοια θα μεταφερθούν σε δημοτικό επίπεδο, σε επίπεδο δήμων και δημιουργούνται προπαρασκευαστικές ε, ομάδες για την δημιουργία πέντε νέων δήμων ε, μέχρι το τέλος του Μαρτίου. Γίνονται προσπάθειες μεταρρύθμιση τομέα της παιδείας και κατάρτιση προγράμματος, σχολικού προγράμματος για τα σερβικά σχολεία που επίσης ελπίζουμε να ολοκληρωθούν αυτές τις προσπάθειες μέχρι το τέλος ε, Μαρτίου. Κύριε Πρόεδρε, οι ανησυχίες που εκφράσατε στο ψήφισμά σας σχετικά με την επιστροφή των μειονοτήτων και των εκτοπιστέντων ε, είναι ανησυχίες που ενστερνίζομαι και εγώ και συνεχώς ασχολούμεθα με αυτά τα θέματα και το συζητούμε το ζήτημα αυτό με τις αρχές. Το Υπουργείο Κοινοτήτων και Επιστροφών Επαναπατρισμών σε συνεργασία με το UNDP και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, θα υποστηρίξουν τη διαδικασία επιστροφής των διαφόρων πολιτών και διέθεσε περαιτέρω πόρους στο αρμόδιο Υπουργείο για την παιδεία, για τη στέγαση των κοινοτήτων και για την επιστροφή των ανθρώπων στις διάφορες κοινότητες. Παρόλο που η διαθέσιμη πόρη είναι μέτρη, η κυβέρνηση είχε δεσμευθεί να εργαστεί άοκνα στον τομέα αυτό. Αρκετές προκλήσεις εκρεμούν, πρέπει να δημιουργηθεί το κατάλληλο περιβάλλον για αυξημένες ροές επιστροφών και ένταξη των μειονοτικών κοινοτήτων στην καθημερινή ζωή του κοσυφοπεδίου. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας ώστε να καλύψουμε αυτά τα ζητήματα σε στενή συνεργασία με τις αρχές. Κυρίες και κύριοι, όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα της κοινότητας των Ρώμα, που έχει πληγεί από δηλητηρίαση από μόλιβδο ε, στο βόρειο υποπέδιο. είμαι ικανοποιημένο διότι ακολουθεί τη σωστή διαδικασία για να κλείσουν τα ε, στατόπεδα εκεί οι κατασκηνώσεις εκεί και οι Ρώμα να πάνε σε ασφαλείς περιοχές με πολύ καλή, καλές συνθήκες, ε, συνθήκες. Αυτή η διαδικασία παρεμποδίζεται τώρα λόγω έλλειψης επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων φορέων στο βορρά και στο νότο. Και είναι ασταθής η πολιτική κατάσταση στην, στο βορρά της, του Κωσυφοπεδίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με το αρμόδιο γραφείο της στην Πριστίνα, συντονίζει τους προσπάθειες εθνικών και διεθνών φορέων ούτως ώστε να εξευρεθούν μακροπρόθεσμες βιώσιμες λύσεις. Κύριε Πρόεδρε, εν κατακλείδη, φιλόδοξο πρόγραμμα μας περιμένει για το κοσυφοπέδιο, Περιμένει τη διεθνή κοινότητα και κυρίως την Ευρωπαϊκή Ένωση το επόμενο έτος. Αλλά με επαρκή πολιτική βούληση, με συντονισμό και ενθάρρυνση η κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου θα μπορέσει να σημειώσει πρόοδο όσον αφορά την ευρωπαϊκή της πορεία. Από αυτά που είπα Υπάρχουν πολλές αποδείξεις ότι οι διπλές μου ευθύνε στο κοσυφοπέδιο έχουν αυξηθεί ε, συμπληρώνοντας η μία την άλλη και μπορώ να συνομιλώ με διάφορες πλευρές έχοντας το κατάλληλο κύρος και με μεγαλύτερη πιθανότητα επιτεύξεως των τεθέντων στόχων. Θα ήθελα για μία ακόμη φορά να σας ευχαριστήσω για την υποστήριξή σας και για το ισχυρό ψήφισμα που προσέθεσε ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό και ορμή στην ομάδα μου και σε μένα στις προσπάθειες που καταβάλουμε για να βοηθήσουμε το λαό του Κωσυφοπεδίου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ κύριε εκπρόσωπε. Καλύψατε ένα ευρύτερο φάσμα θεμάτων. Να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο πρώτος είναι ο εισηγητής, ο κύριος Λάγκεντακ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, είχα τη δυνατότητα να μεταβώ στο κοσυφοπέδιο, αμέσως μετά την ψηφοφορία μας την περασμένη Πέμπτη. Πέρασα λοιπόν το Σαββατοκύριακό μου στην Πρίστανα και έκανα και μια περιοδία στο κοσυφοπέδιο και θα ήθελα να σας δώσω λίγο τις εντυπώσεις μου από το ταξίδι αυτό. Η έκθεσή μας ε, έχει λάβει θετικά σχόλια όχι μόνο από εμά αλλά και από τους εκπροσώπους της διεθνούς κοινότητας όπως ε, επεσήμανε και ο ειδικό εκπρόσωπος και ήταν ευχάριστο το γεγονός ότι επιτέλους η Ulox κατάφερε να ε, να αναπτυχθεί σε όλη την ε, επικράτεια του Κωσυφοπεδίου. Μίλησα με τη Γιουλόπ και με το προσωπικό του ICO επιτόπου, με τελωνιακούς υπαλλήλου, ε, με αστυνομικούς, ε, με δικαστές ε, και νομίζω ότι έχουν καταφέρει να λάβουν, να συνδυάσουν όλα αυτά τα που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε στο κοσυφοπαίδιο. Διπλωματικές δεξιότητες, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και υπομονή. Και εξεπλάγει με ευχάριστο τρόπο ε, διαπιστώνοντας ότι το έργο των δικαστών ε, των ε, τελωνιακών υπολογιών πολλές φορές παρακολύεται από το γεγονός ότι δεν έχουν εξοπλισμό, δεν έχουν δυνατότητες πληροφορικής που υποσκάπτει όλες τις ενέργειες αυτών των ανθρώπων που ουσιαστικά θέλουν να βοηθήσουν το κοσυποπέδιο και η Ευρωπαϊκή Αποστολή ορισμένες φορές δυσκολεύεται. Ορισμένες φορές έχουμε καθυστερήσεις ακόμα και από διαδικασίες προμηθειών εδώ στις Βρυξέλλες, όχι από τους ανθρώπους που βρίσκονται επί τόπου, αλλά με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε διευθετήσει εμείς τις δουλειές μας εδώ, το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι κρίμα να παρακολύεται το έργο τους από ε, τέτοια προσκόμματα και νομίζω ότι αυτό θα το ε, ήθελα να το λάβουμε υπόψη μας σε σχέση μας με την ε, επαφές μας με το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε με κάποιο τρόπο να το βγάλουμε από τη μέση. Αυτό που επεσήμανε επίσης και ο ειδικό εκπρόσωπος στην ομιλία του είναι το γεγονός που μας επεσήμαναν και όλοι όσοι με τους οποίους μιλήσαμε στην αποστολή μας στο Κωσυφοπέδιο. Αυτή η αποστολή μπορεί να επιτύχει μόνο αν υπάρχει επαρκή συνεργασία μεταξύ της ULEX και των σερβικών αρχών στο Βελιγράδο η συμμετοχή των ε, Σέρβων του Κωσόβου στο, ε, στα τοπικά συμβούλια και, στα εθνικά, και στις εθνικούς φορείς είναι πάρα πολύ σημαντική και δείχνει ότι θέλουν και αυτοί να συμμετέχουν, αλλά θα το κάνουν μαζικά εάν λάβουν ένα πράσινο φως από τη Σερβία και όχι το κόκκινο φως που λαμβάνουν αυτή τη στιγμή και τους λέει ότι ε, δεν θα έπρεπε να συμμετέχουν αν ε, θέλουν και να είναι πιο μέτρια η συμμετοχή τους. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι πάρα πολύ αποκρισταλωμένο στο μήνυμα που θα αποστείλουμε στο Βελιγράδι. Το έχω πει και επανειλημμένω, δεν μου αρέσει ούτε καν η πολιτική τη δική μου χώρα που δυσχεραίνει τη ζωή του Βελιγραδίου και δεν επιτρέπει και την προσέγγιση Ευρωπαϊκή Ένωση Σερβία. Πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα, αλλά αυτά μπορούν να γίνουν μόνο όταν υπάρχει σαφή συνεργασία από το Βελιγράδι και υπάρχει και ε, η αίσθηση ότι το να επιτρέπουμε την παρουσία του γιουλέξου στους δικαστές, στους αστυνομικούς ε, να κάνουν τη δουλειά τους, ε, αυτό είναι ικανή και αναγκαία συνθήκη. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόοδο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Σερβίας εάν το Βελιγράδι δημιουργεί προβλήματα στους ανθρώπους μας, κυρίως προς το βορρά. Αυτό το μήνυμα θα πρέπει να αποσταλεί σαφέστατα και ε, νομίζω ότι το Βελιγράδι θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η επιτυχία αυτής της αποστολής θα πρέπει να εξαρτάται και από αυτούς. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, το κατάλαβα και από τους ανθρώπους με τους οποίους μίλησα επί τόπου. Και αυτό ε, νομίζω ότι θα προκύψει και από τις μελλοντικέ συζητήσεις που θα κάνουμε για το Κωσυφοπέδιο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Πάκα, ευχαριστώ πολύ κύριε Φάιτ. Καλώς ήλθατε. χωρίς καμία μετάβαση μπορώ να υποστηρίξω αυτά τα οποία είπε ο κύριος Λάγεντάικ. Νομίζω ότι το έργο της ε, EULEX κάνει μια πραγματικά ποιοτική διαφορά σε σχέση με το έργο της UNMIC. Αυτό για να είναι πραγματικότητα πρέπει να εξασφαλίσουμε την καλή ποιότητα της εργασίας της EULEX. Έχουμε πολλά άτομα τα οποία είναι πραγματικά υψηλών προσόντων και που θα δώσουν τη δυνατότητα σε αυτούς οι οποίοι ζουν στο Κόσοβο να μεταρρυθμίσουν τη χώρα τους. Πρέπει να υποστηρίξουμε όλη την Ulex και εμείς αναγνωρίσουμε όλοι ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά χρειάζεται και η υποστήριξη του Βελιγραδίου. Υπάρχει πραγματικά μεγάλη προσδοκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση των πολιτών του Κωσυφοπεδίου, αλλά εμείς θα πρέπει σε όλες τις περιπτώσεις που ερχόμαστε σε επαφή με το Βελιγράδι να τονίσουμε το ενδιαφέρον μας για την επίτευξη μια σταθερότητα και ευμάρεια στο κοσμοπέδιο. Δεν μπορούμε να παραγνωρίσουμε το θέμα αυτό. Το Βελιγράδι ζητά να γίνει μια χώρα, η Σερβία, μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να του πούμε όμω ότι για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει να βοηθήσετε ώστε οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν σε μια γειτονική τη χώρα να ζουν σε ένα επίπεδο ομαλότο. Και αυτό περιλαμβάνει και πολλού Σέρβου, όχι μόνο στη Μητρόβιτσα, αλλά σε όλη την ε, <clears throat> επικράτεια του κοσμοπεδίου και όχι μόνο στο βορρά. Εγώ λοιπόν θα χαιρόμουν πάρα πολύ για το γεγονός ότι θα αν προχωρήσουν πραγματικά οι στρογγυλές τράπεζες όχι μόνο για την υγειονομική περίθαλψη αλλά και για τα θέματα της εκπαίδευσης. Και πράγματι είναι καιρός εμείς να παίξουμε κάποιο ρόλο στα θέματα αυτά μετά από τα 10 χρόνια που είμαστε εκεί. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι σωστή η προσέγγιση της Ulex αλλά υπάρχει κι άλλο ένα πρόβλημα το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε σχέση με τα γειτονικά κράτη. Υπάρχουν πολλέ περιπτώσει οι οποίε παραμένουν ακόμα εκρεμή σε επίπεδο δικαστική δίωξη. Θα πρέπει να προχωρήσουν όλα αυτά. Είναι πάρα πολλέ οι περιπτώσει ατόμων για τα οποία έχουν απαγγελθεί κατά κατηγορία αλλά δεν έχουν έρθει ενώπιον των δικαστηρίων ακόμα και αυτό δηλητηριάζει το κλίμα στο κοσυφοπαίδιο. Δεν νομίζω ότι αυτό έχει γίνει λόγω κακής θέλησης, αλλά ήταν μια έλλειψη οργάνωσης. Γι' αυτό ελπίζω ότι η EULEX θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Επίσης έρχομαι στο θέμα των τοπικών εκλογών, των δημοτικών εκλογών. Κατανοώ ότι δεν μπορούν να γίνουν εφέτος οι εκλογές αυτές, δεν είναι μια μεγάλη απώλεια. Πρέπει πρώτα να υπάρξει μια πραγματική ε, οργάνωση του κράτους του φτάσουμε σε γενικές εκλογές. Αλλά για τις τοπικές εκλογές νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο να γίνει. Το προέβλεπε και το σχέδιο Αχτισάρι να έχουμε μια πραγματική αποκέντρωση στο κοσμοπέδιο. Είναι απαραίτητο λοιπόν να γίνουν αυτές οι εκλογές ώστε οι νέες αυτές τοπικές και περιφερειακές διαιρέσεις του κοσφοπεδίου να μπορέσουν να έχουν την απαραίτητη αυτονομία τους και να εκλέξουν τους τοπικούς αρχηγούς λαμβάνοντας υπόψη και την αυθινοτική σύνθεσή τους. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρέπει να προωθήσουμε με έντονο τρόπο την αποκέντρωση γιατί αυτό είναι προϋπόθεση για να υπάρξουν και οι εκλογές στο επίπεδο αυτό. Επίσης είναι σημαντικό να δώσουμε προοπτική στους νέους στο κοσμοπέδιο να έχουν μια επαφή μεταξύ τους ανεξάρτητα από την εθνοτική τους προέλευση, να έχουν επαφές με τους ε, <clears throat> άλλους λαούς της περιοχής πέραν της Μετρόβιτσα, πέραν της Πρίστινα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα να υπάρξει ένα ευρωπαϊκό ανώτατο ίδρυμα στο οποίο θα μπορούν όλοι να εργάζονται και να μαθαίνουν ίσως σε μια κοινή γλώσσα που θα είναι τα αγγλικά σε μια ευρωπαϊκή γλώσσα. Εσείς κύριε Φέιτ ξέρετε ότι θα μπορούσατε να έχετε μια τέτοια δομή πανεπιστημιακή στο οπότε θα έχετε και ένα φάρο ο οποίος θα προσελκύσει και ανθρώπους από τη Μακεδονία, από τα άλλα κράματα της περιοχής. Πιστεύω λοιπόν ότι αν προχωρήσετε με τις πρωτοβουλίες των στρογγυλών τραπεζών στο κοσφοπέδιο και υπάρξει και συνεργασία μεταξύ τους, μπορούμε να επιτύχουμε μια δέσμευση όλου για, ένα συνολική, για μια συνολική αντιμετώπιση στο Κωσυφοπέδιο. Ευχαριστώ κύριε Πακ και ήθελα κύριο Σφόμοντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Φάιντ για την παρουσίασή του που μας έδωσε. Έχει και θετικά στοιχεία βέβαια και αντικά στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση στο κοσυφοπέδιο. Θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα σημεία. Καταρχήν εμείς είμαστε κοινοβουλευτικοί και επομένως είναι απαραίτητο από το δικό μας κοινοβούλιο να σας υποστηρίξουμε με το μήνυμα ότι πρέπει να λειτουργήσει και το κοσφοπέδιο στο κοσφοπέδιο. Είναι το κέντρο της δημοκρατίας. Δεν μπορούν οι αποφάσεις να λαμβάνονται μόνο από μια κυβέρνηση, αλλά και από ένα κοινοβούλιο το οποίο λειτουργεί με ομαλό τρόπο. Αυτό δίνει και περισσότερες δυνατότητες να υπάρξει μια ολοκλήρωση μεταξύ των διαφόρων ομάδων όταν υπάρχει η ευκαιρία σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να ανταλλάσσουν απόψεις και να συναποφασίζουν. Τώρα το δεύμα των εθνοτικών ομάδων, ιδίως των Σέρβων. Όπως είπε και η Doris Park, η Doris Ξέρουμε ότι υπάρχουν περιοχές και τομείς όπου συμμετέχουν και οι εκπρόσωποι του Βορρά, δηλαδή οι Σέρβοι. Αλλά το θέμα είναι να μπορέσουν να προχωρήσουν σε πιο συγκεκριμένο επίπεδο. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είπε ο Ιωσ Λάγκεντακ ότι το Βελιγράδι θα πρέπει να δώσει ένα πράσινο φως ή τουλάχιστον να αποσύρει το κόκκινο φως για τη συνεργασία των Σέρβων στο Κωσικοπαίδιο. Το πιο σημαντικό όμως είναι να μπορούν οι άνθρωποι επιτοπίως να συζητούν με τους ε, συμπολίτε του από άλλε εθνότητε και να βρίσκουν λύσει. Μέσα στα πλαίσια αυτά το θέμα των τοπικών εκλογών βέβαια θα ήταν καλύτερο πρώτα να γίνουν οι απαραίτητε μεταρρυθμίσει αλλά από την άλλη πλευρά για μένα μου φαίνεται πάρα πολύ σημαντικό ότι οι τοπικέ εκλογέ θα συμβάλλουν και στην ολοκλήρωση των Σέρβων και των άλλων μειονοτήτων μέσα στο Κοσμοπέδιο. Θα υπάρξει δυνατότητα λοιπόν για αυτές τις μικρότερες εθνοτικές ομάδες να έχουν και μια επιρροή σε τοπικό επίπεδο. Θα μπορούν λοιπόν έτσι να επηρεάσουν περισσότερο την κοινή πορεία του Κοσμοπέδιου. Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να έχει επιτευχθεί όλη η μεταρρύθμιση και η αποκέντρωση. Απλώς να εξασφαλίσουμε ότι όταν θα γίνουν οι τοπικές εκλογές αυτό θα οδηγήσει σε κατακαιρματισμό αλλά σε περισσότερη ενότητα. Και τέλος το θέμα της κατάστασης στο Ρώμα και η περιοχή όπου υπάρξει, έχει υπάρξει δηλητηρίαση από τα μεταλλεία. Εμείς ήδη έχουμε κάνει αυτές τις συζητήσεις μαζί και με την Doris Πακ μέσα στα πλαίσια της διακοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας έχουμε μιλήσει εκεί με τους τοπικούς εκπροσώπους και τους ε, έχουμε ζητήσει να αντιμετωπίσουν τα θέματα αυτής της ε, μειονότητος, ιδίως σε ό,τι αφορά τα προβλήματα υγείας που έχουν ε, παρουσιαστεί στην περιοχή αυτή. Βλέπουμε ότι ολόκληρε γενιέ έχουν θυγεί από αυτό το πρόβλημα. Βλέπουμε πολλέ φορέ ότι είναι καταστροφική κατάσταση στα πιο ηλικιωμένα άτομα, αλλά είναι ακόμα και παιδιά τα οποία έχουν πληγεί από αυτή την δηλητηρία και θέλω να ευχαριστήσω τον εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το έργο του στο Κωσυφοπέδιο. Η ε, κυρία Μπισάτσετς έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. ευχαριστούμε που ήρθατε να μας παρουσιάσετε την έκθεση. Συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση σας σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στο κοσυφοπέδιο αναφερθήκατε σε μια πρώτη συνάντηση, σε μια πρώτη συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των διαφόρων κοινοτήτων που έλαβε χώρα και είχε θέμα τη διατήρηση της κληρονομιάς. Είναι σημαντικό να ε, διατηρηθεί και η κληρονομιά που έχει προστατευτεί από, τις από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Πολύ συχνά όμως το Βελιγράδι αρνείται τέτοιου είδου συναντήσει. Πρέπει να προστατευτεί η κληρονομιά, να διατηρηθεί ούτω ώστε ο καθένα να μπορεί να τη γνωρίσει και οι κοινότητε να μπορούν να συμβιώνουν. Έχετε προβλέψει κάποια προγράμματα για να ενθαρρύνετε τη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς. Έχετε πρόθεση να διαδραματίσετε ένα ρόλο στην διατήρηση αυτής της κληρονομιάς, στη συντήρηση της και ε, την ενημέρωση της κοινή γνώμης. Πολύ συχνά διαπιστώνεται ότι δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη μόνο η γειτονία των χωρών. Θα πρέπει οι άνθρωποι εντός της χώρας να μάθουν τι είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να μάθουν σε αυτές τις χώρες ποιες είναι οι ευρωπαϊκές χώρες. Εξού και το ερώτημά μου. Έχετε εξετάσει το ενδεχόμενο να λάβετε σχετική πρωτοβουλία συγκρίσιμη με αυτό που κάνουν οι εκπρόσωποι μας την έκαναν στη Βοσνία. Ευχαριστώ κύριος Πρίμπετιτς έχει το λόγο σας, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να χαιρετήσω τον ε, συγκητή τον κύριο που έδωσε, μας παρουσίασε το όραμά του και έκανε συστάσεις για να τροφοδοτήσει η συζήτηση μας. Έχω ένα πρόβλημα όσον αφορά την όλη αξιολόγηση της καταστάσεως και έχω την εντύπωση ότι κάνουμε ένα ε, πολύ δύσκολο διάβημα που θυμίζει Κάφκα. Η Σερβία δεν αναγνωρίζει το κοσυφοπέδιο, επουδενή δεν αναγνωρίζει αυτό που θεωρεί ότι είναι παραβίαση των εθνικών της δικαιωμάτων και μόνο το 1244 Συμβουλίου Ασφαλείας το ψήφισμα αναγνωρίζει για τη Σερβία ότι το κοσυφοπέδιο παραμένει επαρχία της. Πώς θα καταφέρουμε λοιπόν να αλλάξει η κατάσταση εάν επιβάλλουμε στους Σέρβους μια κατάσταση που δεν την επιθυμούν. Ε, και η Κύπρος, η Ισπανία, η Ελλάδα, η Σλοβακία, η Ρουμανία δεν έχουν αναγνωρίσει το κοσυφοπαίδιο. Πώς να νομιμοποιήσουμε αυτή την παραβίαση. Ενώ έχουν ευθύνε αυτές οι χώρες, ίσως λόγω αλληλεγγύης, ίσως ε, και λόγω αρνήσεως να δημιουργηθεί ένα προηγούμενο που δημιουργεί κινδύνους απόσχησης. Μηχανικός πώς ε, τελικά έχουμε, δημιουργούμε ένα φαύλο κύκλο. Ε, δημιουργούνται οι δυνάμεις ασφαλής κοσοφεδίου που δυσαρεστούν τους Σέρβους. Ο κ. Ζέρεμιτς αυτό το φορέα τον θεωρεί παραστατητικό και παράνομο της δυνάμεις ασφαλείας, θεωρεί ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη και ας άμει συμβαίνει τίποτα σε κατάσταση ονειρική εξακολουθεί η διαδικασία χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί χωρίς τους Σέρβους. Δεν ενοχλούνται μόνο οι Σέρβοι, ενοχλούνται από πίσω τους Σέρβους και οι Ρώσοι. Οπότε σταδιακά, προοδευτικά, γίνεται σαν μια χημική αντίδραση. Πλησιάζουμε την δημιουργία TNT, εκρηκτικού, τρινιτροτολουόλης. Ο υπουργό επιφωτισμένο, ο Μπογκδάνοβιτ, επιφωτισμένο του Κωσυφοπέδιου, έλεγε σε μια δήλωσή του ότι θεωρούσε ότι υπήρχαν περίπου 300.000 με παράνομα όπλα εντό του Κωσυφοπέδιου. Και εμεί συνεχίζουμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Να στο δοκαμιλίζουμε. Να συνεχίζουμε μηχανικά, σαν να είναι χώρα, κράτο. Τον Ιούνιο πήγα εκ μέρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανα μια αποστολή εκεί για έλεγχο προπολογισμού. Πήγα στο, στη μονάδα παραγωγή τη Πριστίνα, παραγωγή ενέργεια, δεν έχουν πληρωθεί λογαριασμοί. Ρώτησα τον Υπουργό, εφόσον είστε υπεύθυνο, θα ζητήσετε τι καθυστερήσει πληρωμών που είναι 300 εκατομμύρια ευρώ που θα είναι χρήσιμο για τη χώρα για να αποκατασταθούν οι ζημίε και να πάτε προμήθειε, θα κάνετε κάποιε για να μπορέσετε να βρεθείτε σε μια κατάσταση υπευθυνότητα. Και εμένα αυτή η κατάσταση με ανησυχεί. Με ανησυχεί. Διότι έχουμε δίπλα και τη Μακεδονία, έχουμε και άλλα στοιχεία και υπάρχει γενικός οικονομικός μαρασμός. Πώς αυτή η χώρα που αναγνωρίσαμε εμείς θα μπορέσει οικονομικός πώς να βρει τα μέσα για να αναπτυχθεί ενώ η Σερβία δεν θέλει να συμμετάσχει στη διαδικασία και δεν θα συμμετάσχει. Λοιπόν, εγώ έχω ένα σχόλιο επί της ουσίας όσον αφορά την αντίληψη των πραγμάτων, την προσέγγιση των πραγμάτων και την εθελοτυφλία μας όσον αφορά την κατάσταση. Λοιπόν, ξεκίσαμε τι ήθελε να κάνει ο Τίτο, να κατοικείται το Κωσοπέδιο από Αλβανόφωνος για να υλοποιηθεί και το όνειρο τελικά της ε, Μεγάλης Αλβανίας. Ευχαριστώ. Δίνω το λόγο τώρα στον κύριο Φέιθ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Um, να απαντήσω σε κάποια από τα θέματα που αναφέρατε σε αυτό τον πρώτο γύρο, αλλά πριν από αυτό να κάνω ένα γενικό σχόλιο. Δεν είμαι επικεφαλής της αποστολής της EULEX. Ο στρατηγός Δεκαμαμπό είναι υπεύθυνος για το EULEX Έχω πολύ καλή σχέση με τον στρατηγό. διότι έχω λάβει και εντολή από το Συμβούλιο για τοπική πολιτική καθοδήγηση. Και όπως αυτό το έχει αναγνωρίσει και το ψήφισμά σας, η αποστολή θα πρέπει να συνεργάζεται στενά με τη δική μου ομάδα. Και αυτό συμβαίνει. Θα πρέπει βέβαια να σας προειδοποιήσω ότι ο στρατηγός Καμαμπό δεν θα ήταν χαρούμενος αν προσπαθήσω εγώ να απαντήσω κάποια από τα επιχειρησιακά θέματα που μου θέσατε. Αυτό που θα κάνω είναι να του μεταφέρω τις παρατηρήσεις σας και να του ζητήσω να δώσει τη δέουσα προσοχή στις ανησυχίες σας. Θα πρέπει όμως να επαναλάβω εξ του ότι η ανάπτυξη στο Κωσυφοπαίδιο από το Δεκέμβριο και τούδε είναι κάτι το οποίο έχει αναγνωρίσει ευρέω ε, ο λαός του Κωσυφοπαίδιου ως επιτυχία, ως ένα καλό πρωτοβήμα και μια ευπρόσδεκτη εξέλιξη σε σχέση με την ε, αποστολή των Ηνωμένων Εθνών στο Κωσυφοπαίδιο και το πώς εξελίχθηκε και ο κόσμος περιμένει με ανυπομονησία την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει η EULEX. Δεύτερη παρατήρηση. Ο διάλογος με τις κοινότητες και κυρίως τους Σέρβους εκπροσώπους. Μπορούν να γίνουν πολλά. και πολλοί από τους ε, Σέρβους ηγέτες του Κωσυφοπεδίου επιδεικνύουν ιδιαίτερο θάρρος και είναι διατεθειμένοι να ξεκινήσει αυτός ο διάλογος. Δεν πρόκειται για ένα διάλογο ο οποίος θα γίνεται μεταξύ αυτών και μου. Εγώ θέλω να κάτσουν σε ένα τραπέζι, να ξέρω ότι θα υπάρχει καφές και νερό και είναι ένας διάλογος ο οποίος θα πρέπει να ξεκινήσει με τους εκπροσώπους της κυβέρνησης στην Πρίστινα. Να σας πω όμως ότι οι Σέρβοι εκπρόσωποι ε, ένιωσαν καλά, πήραν θάρρος από αυτή την πρώτη συνάντηση με την ε, κυβέρνηση του Κωσυφοπεδίου και είναι διατεθειμένοι να συνεργαστούν. Αλλά, όπως είπατε και εσείς, θα βοηθήσει τα μάλλα να λάβουν περισσότερη ενθάρρυνση από ε, το Βελιγράδι. Πρόκειται για μια ευρωπαϊκή αρχή, την οποία πάντα επαναλαμβάνω σε όσους ε, με παρακολουθούν στο ακροατήριό μου στο Κωσυφοπαίδιο. Είναι μια πολυεθνική κοινωνία, πρέπει να συμβιώσουν, υπάρχουν δυνατότητες που εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να τους παράσχουμε, και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση δεν υποστηρίζουμε την ε, άρση τυχών και την ε, δημιουργία χασμάτων μεταξύ των διαφόρων εθνικών, ε, εθνοτικών κοινοτήτων. Θεωρώ ότι αυτό το μήνυμα σταδιακά γίνεται κατανοητό στο κοσφοπέδιο και πιστεύω ότι θα περάσει το ίδιο μήνυμα και στο Βελιγράδι. Τελικά. να αναφερθώ κυρίως στην πολιτιστική και θρησκευτική κληρονομιά σε αυτό το πλαίσιο. Η άποψή μου και πάλι είναι ότι αν θέλουμε να έχουμε μια βιώσιμη λύση που θα προστατεύσει τα σερβικά μνημεία, της εκκλησίες τους, καθώς και τα μνημεία των άλλων κοινοτήτων, δεν υπάρχει έλα εναλλακτική λύση. Ε, η μόνη εναλλακτική λύση είναι η πλήρη συνεργασία των ε, κοινοτήτων. Εμείς μπορούμε να δίνουμε συνεχώς στρατιώτες ε, να φιλούν τα σέρβικα μοναστήρια στο Κοσφοπέδιο, αλλά ειλικρινά πρέπει να σας πω ότι δεν τους έχουμε γι' αυτό τους στρατιώτες. Ο στρατός μας θα πρέπει να αναπτυχθεί και να μπορέσει να ασχοληθεί με άλλα καθήκοντα. Επομένως, η βιώσιμη λύση είναι η αστυνομία του Κωσυφοπεδίου, που τώρα χάρη στις προσπάθειες των Ηνωμένων Εθνών τα τελευταία 9 χρόνια έχει φτάσει σε ένα επίπεδο επαγγελματικό αξιοσημείωτο. Θα πρέπει λοιπόν αυτοί να αναλάβουν αυτές, αυτά τα καθήκοντα. Και θεωρώ ότι για το μέλλον αυτή είναι η κατεύθυνση που θα πρέπει να ακολουθήσουμε στόχος μου είναι να μαζευτούν οι τοπικές αρχές με εκπροσώπους της Σερβικής Κυβέρνησης και της Σερβικής Ορθόδοξης Εκκλησίας και θα τους ζητήσω να ε, θεωρήσουν ως κάτι θετικό τη συμμετοχή σε αυτή την προσπάθεια, διότι αλλιώς χρονοτριβούμε και ίσως ε, η κατάσταση μπορεί να οπισθοχωρήσει και πάλι και να έχουμε και νέα προβλήματα. Τώρα για τις δημοτικές εκλογές. είστε ενώπιον ενό ε, διλήμματος. Η ιδανική κατάσταση, και αυτό θα προσπαθήσω να επιτύχω, είναι να καθοριστεί ε, το πότε θα γίνουν ε, σε σχέση με την πρόοδο για την αποκέντρωση και αυτό θα το δούμε και στις επαφές μας με την σέρβικη κοινότητα του Κοσφοπεδίου. Κανονικά θα πρέπει να γίνουν ε, στο τέλος του χρόνου, διότι τότε θα έχει παρελθεί το διάστημα των δύο ετών. Αν όμως δεν υπάρχει επαρκής πρόοδος μέχρι τότε, θα κάνω ό,τι μπορώ και θα λάβω υπόψη μου και το σχόλιο της κυρίας Πακ νομίζω, ότι αυτός είναι ένας λόγος παραπάνω για να πιέσουμε ακόμα περισσότερο το θέμα της αποκέντρωσης και αυτό θα κάνουμε. Σε γενικές γραμμές όμως, και αυτό Ίσως είναι κάτι το οποίο θα ήθελα να ζητήσω από τον κύριο Πρίμπετης να λάβει υπόψη του. Άκουσα την ανάλυση σας. Αλλά νομίζω ότι το συμπέρασμα δεν μπορεί να είναι ότι τα πάντα εξαρτώνται από το Βελιγράδι και τους Σέρβους του Κωσυφοπεδίου. Δεν μπορούμε, για χάρη της σταθερότητας ε, στα Βαλκάνια, να θέσουμε βέτο στην ε, κοινότητα των Σέρβων ε, στο Κωσυφοπαίδιο και στους Σέρβους. Ε, δεν το υπαγορεύει λογική σε καμία περίπτωση αυτό, δεν μπορούμε να διατηρήσουμε τη σταθερότητα βάση αυτού και φρονώ ότι θα μας κάνει να χάσουμε και το στόχο μας για τις ευρωπαϊκές προοπτικές που έχουμε δώσει στη Σερβία και στο Κωσυφοπαίδιο. Βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύ περίπλοκης κατάστασης, συμφωνώ μαζί σας, θα ήταν ευσεβής πόθος να ήταν πολύ καλύτερη κατάσταση από πολλές ε, πλευρές. Ε, θα μπορούσαμε να είχαμε ξεκινήσει από μια ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό θα ήταν σίγουρα καλύτερο. Δυστυχώς όμως, κύριε Πρόεδρε, δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Δεν συμφώνησαν τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, αλλά η οπλή ψηφία των χωρών ε, που εργάζονται στο θέμα των Βαλκανίων κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική λύση πέραν της ανεξαρτησίας. Γι' αυτό λοιπόν αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προχωρήσουμε. Έχουμε μια απόφαση του Συμβουλίου την οποία γνωρίζετε, ε, ελήφθη στις αρχές του περασμένου έτους και δίνει στο κοσφοπέδιο τη δυνατότητα για μια αποστολή κράτους δικαίου. Δεν μπορούμε να μιλάμε για όφελος εδώ, αλλά θα υπάρχει τέλος πάντων ένα διεθνές ε, γραφείο παρακολούθησης. Όλα αυτά είναι μέσα για να βοηθήσουμε το λαό του Κοσφοποδίου να προχωρήσει και να έχει ένα πολυεθνικό και βιώσιμο περιβάλλον. Και παρά το γεγονός ότι συμφωνώ μαζί σας ότι Υπάρχουν δύσκολες προκλήσεις, όπως για παράδειγμα αναφέρατε το θέμα της, ε, των δυνάμεων ασφαλείας του κοσυφοπεδίου θα το, ε, θα το προσπαθήσουμε αυτό το θέμα, διότι θεωρούμε ότι είναι καλύτερα να έχουμε δυνάμεις ασφαλείας ε, εθνικού ελέγχου, έστω και μικρές, παρά να έχουμε παραστρατιωτικές παράνομες ομάδες που θα αναπτυχθούν στο κοσφοπέδιο και θα δημιουργούν προβλήματα. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό είναι πρόοδος. Μπορεί εσείς να βγάζετε διαφορετικό συμπέρασμα, αλλά το συμπέρασμα είναι ότι αυτά τα οποία θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για 2.000 ε, άντρες, δεν ε, θα είναι τεράστια αυτή η δύναμη, αλλά αυτό που θα κάνουν θα είναι κυρίως υποστήριξη του πληθυσμού σε περιόδους εθνικών καταστροφών και νομίζω ότι πρόκειται για ένα θετικό βήμα. Δεν συμφωνώ μαζί σας ως προς τον κίνδυνο της δημιουργίας μιας ευρύτερης Αλβανίας. Εγώ συμφωνώ με τα συμπεράσματα της ομάδας επαφής συμπεριλαμβανομένους και της Ρωσίας και των πέντε δυτικών εταίρων ότι υπάρχουν κάποιες αρχές οι οποίες θα πρέπει να γίνονται σεβαστές όταν ε, εξετάζουμε την περαιτέρω κατάστασή τους και αυτό, μία εξ αυτών είναι ότι δεν υπάρχει κανένας διαχωρισμός και δεύτερον το κοσφοπέδιο δεν θα ενωθεί με μία από τις γείτονες χώρες. Νομίζω ότι αυτό είναι δεδομένο και δεν βλέπω καμία ένδειξη αυτή τη στιγμή και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει καμία τέτοια εξέλιξη. Ε, δεν ε, θα ε, ενταχθεί το κοσφοπέδιο στην ευρύτερη Αλβανία. Uh, Ευχαριστούμε κύριε Φέιτ για αυτό το πρώτο γύρο συζητήσεων και ο κύριος Μέγιας για το δεύτερο. Voorzitter, Een ε, Πρόεδρε. Μια σημαντική παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο κοσμοπέδιο μπορεί να ενδιαφέρουσε για πολλούς λόγους. Πρώτον, από τη μεταβατική περίοδο από τον περασμένο Ιανουάριο, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους δηλαδή, θα μπορούσε να αποφύγει το, την εφαρμογή του χάους. Και νομίζω ότι η περίοδος αυτή θα εμφανίστηκαν στο ξεκίνημα, αλλά οι συνέπειές της τώρα διαπιστώνονται. Η εγκατάσταση, η επιστροφή μάλλον των Ρωμά είναι βασικό στοιχείο για να διαπιστώσουμε κατά πόσον δεν θα υπάρχουν ε, διακρίσεις και ότι όλες οι ομάδες μπορούν και έχουν δυνατότητα να ενταχθούν. Κατόπιν, διοίκηση. Ο στόχος δεν είναι να υπάρχει πραγματική παρέμβαση. Το είδαμε στη Βοσνία αυτό. Αλλά να προσφέρουμε ποιότητα και συμβουλές ποιότητας. Επίσης, διαπιστώνω ότι στο Κωσυφοπέδιο υπάρχει ο φόβος ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αρχίσει να εμπλέκεται στις εσωτερικές υποθέσεις τους. Όλα αυτά, ωστόσο το ευρωπαϊκό μέλλον του Κωσυφοπέδιου παραπέμπεται στο απότερο μέλλον, ενώ ο στόχος μας θα πρέπει να είναι να, προσχωρήσουμε, να προχωρήσουμε ταχύτερα, όσο ταχύτερα γίνεται στην ένταξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το άκουσα στην εισήγηση. Πιστεύω ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Δηλαδή, ο κύριος Φέιτ το είπε με σωστό τρόπο, έχει στόχο, λέει, θέλει μάλλον, να δημιουργήσει μια πολυεθνική κοινωνία. Εγώ είμαι πολύ απεσιόδοξο στο σημείο αυτό. Πιστεύω ότι πρόκειται για πολύ δύσκολο έργο να θέλουμε να κάνουμε το κοσυφοπέδιο μία χωριστή οντότητα. Είναι πολύ αδύνατο. Είναι αδύνατο πραγματικά, εξαιρετικά δύσκολο τουλάχιστον. Το κοσυφοπέδιο σαν ανεξάρτητο είναι ανεξάρτητη χώρα, η πλειοψηφία είναι Αλβανοί, οι οποίοι έκοψαν σχέσεις με την ριζοσπαστική, με τους ριζοσπάστες Σέρβους. Αυτά είναι χαρακτηριστικά που δεν μπορούμε να γνωρούμε. Πιστεύω ότι το να θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα από την άλλη, από μακριά, δημιουργεί εντάσεις και απογοητεύσεις από όλες τις πλευρές. Και από την πλειοψηφία και από αυτούς που βρίσκονται στο βορρά στην Μητρόβιτσα που δεν θέλουν να κόψουν τις σχέσεις τους με την Σερβία και να ε, μπουν στο νέο κράτος, θέλουν να κρατήσουν τη, τα, τελωνία τους, τις δημόσιες υπηρεσίες της Σερβίας και αυτό είναι άποψη της πλειοψηφίας εκεί. Από την άλλη μεριά έχουμε τους νότιους, ε, κυρίως τους Αλβανούς ε, στην περιοχή αυτή όπου οι Σέρβοι είναι μειοψηφία και θέλουν την ένταξη, αλλά οι Αλβανοί θέλουν μια απόλυτη ανεξαρτησία και καμία εποπτεία και επίβλεψη απ' έξω. Ρωτώ λοιπόν κύριε Φάιτ, Πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να συνδιαλέξουμε τις δύο αυτές θέσεις, πλήρη ανεξαρτησία από τη μια μεριά και τους άλλους που θεωρούν ότι πάντοτε είναι Σέρβοι και θέλουν να κρατήσουν στενούς δεσμούς με τη Σερβία. Πότε θα μπορούμε να περιμένουμε αποτελέσματα. Νομίζω ότι πρόκειται για μια αδύναμη, αδύνατη προστασία. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ κύριε Μάιερ, κύριε Γκόμες. Uh, και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Φέιτ για την τόσο εξισορροπημένη παρουσίασή του για την κατάσταση, εξισορροπημένη τουλάχιστον από τη βάση αυτών που γνωρίζω, και να ευχαριστήσω και τον κύριο Λάχεντάικ για την ε, αποστολή παρακολούθησης στην περιοχή και για τα στοιχεία που μας προσέφερε στην παρουσία, στην ομιλία του. Εγώ υποστηρίζω ιδιαίτερα αυτά που έχουν λεχθεί από τον κύριο Φέι, τον κύριο Λάχεντάικ, τον κύριο Σφόμποντα, την κυρία Πακ. Πράγματι θα πρέπει να έχουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια σε σχέση με το Βελιγράδι και αυτό περιλαμβάνει και το κοινοβούλιο μας σε σχέση με το μήνυμα το οποίο περνάμε και σε σχέση με την δράση που περιμένουμε από αυτούς σε σχέση με την κατάσταση στο Βορρά. Όταν μιλάμε για το κοσυφοπέδιο μιλάμε <clears throat> για τις μειονότητες, αλλά μένα με ενδιαφέρουν και οι πλειοψηφίε. Η πλειοψηφία, όπως και σε άλλα μέρη, είναι γυναίκες. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η κατάστασή μας, λοιπόν, σε σχέση με τα δικαιώματα των γυναικών. Έχουμε ένα μεγάλο αριθμό γυναικών στο Κοινοβούλιο <clears throat> που αγωνιστήκαμε να υπάρχουν ποσοστώσεις <clears throat> στο κοινοβούλιο, αλλά λένε ότι πολλές φορές τις παραγνωρίζουν και τις αγνοούν ακόμα και οι εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είπαν ότι σε διπλωματικές θέσεις δεν υπάρχουν καθόλου γυναίκες που έχουν διοριστεί. Στους, στο στρατό επίσης είναι ελάχιστη συμμετοχή των γυναικών, κάπως διαφορετικά τα πράγματα στην αστυνομία. Πού βρίσκεται λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα θέματα αυτά. Έχουμε εστίαση στα θέματα γυναικών στην EULEX, αλλά και πάλι μας λένε ότι δεν τις λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα η EULEX. Και τώρα και πάλι, εν ώψη των, εκλογών που επίκυνται των τοπικών εκλογών, όποτε και να γίνουν, υπάρχει μια διαδικασία που θα εκφράσει την ισότητα ανδρών και γυναικών. Θα υπάρξει ένα σύστημα ισομερές για τη συμμετοχή των γυναικών στις εκλογές και φυσικά και το θέμα της διαφθοράς. Όταν ήμασταν εκεί παρούς, παρόντες στο Κοσμοπέδιο, γυναίκες από το Κοσμοπέδιο, ήταν αυτές οι οργανώσεις τους που είπαν ότι λυπούνται για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η EULEX αναφερόσαν στο θέμα της διαφθοράς και της αντιμετώπισης του οργανωμένου εγκλήματος, αλλά ουσιαστικά κατεφημισμό. Είπαν ότι δεν θα είναι η EU λέξη η θα θέσει αυτό το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ποιο θα το θέσει λοιπόν στη Μέση διάταξη, ποιο θα αντιμετωπίσει τη διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, ποιο θα ζητήσει από τι αρχέ του Κοσφοπεδίου να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα και όχι μονάχα στο βορρά όπου είναι οι τοπικέ σερβικέ ουσιαστικά δυνάμει οι οποίε έχουν την ευθύνη για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριο Ναζάρ. Ευχαριστώ τον κύριο Faith που παρουσίασε πολύ ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες για τις εσωτερικές εξελίξεις του Κωσυφοπαίδιο και θέλω να αναπτυχθεί πολύ καλή σχέση μεταξύ της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κωσυφοπαίδιο και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η χώρα μου δεν αναγνωρίζει βέβαια το Κωσυφοπαίδιο, όμως συμμετέχει με αστυνομικέ δυνάμεις στην εκπροσώπηση Ευρωπαϊκής Ενώσης και ανεξάρτητα από το αν υποστηρίζουμε την εξαρτησία του Κοσμοδίου ή όχι θα πρέπει να συνεργαστούμε ούτως ώστε να είναι σταθερό ε, αυτάρκες και χρειάζεται γι' αυτό ενεργός διάλογος με το Βελιγράδιο και το χρώμα του φωτός που θα δείξει το Βελιγράδιο εξαρτάται την προσέγγιση μας. Η εμπειρία μας δείχνει ότι αποξένωση εδαφική δεν μπορεί να επιβληθεί. Χρειάζεται ρύθμιση με το Βελιγράδι που θα οδηγήσει σε μακροπρόθεσμη σταθερότητα. Παρόλο που παρουσία τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω στο Κωσυφοπαίδιο είναι ευπρόσδεκτη, εγώ δεν θα ήθελα το Κωσυφοπαίδιο να γίνει προτεκτορά τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Θα πρέπει να βοηθήσουμε την Πριστίνα να αναπτύξει του δικού τη θεσμού και τι οικονομικέ δυνατότητε και για αυτόν τον σκοπό θα ήθελα πολύ να ακούσω Ποια είναι η άποψη του κυρίου Φέιθ όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα για την ανάπτυξη της Γιούλεξ στο Κωσυφοπαίδιο. Και το θέτω το ερώτημα γιατί πιστεύω ότι την πρώτη ημέρα θα πρέπει να έχουμε σαφεί προσδοκίε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εντό του οποίου αναμένεται η αποστολή μα να εκπληρώσει του στόχου τη και να επιτρέψουμε στι αρχέ στην Πριστίνα να ε, αναλάβουν πλήρω τα καθήκοντά του όσον αφορά την κυβέρνηση. Βάσει των αντιδράσεων, των συνομιλιών σα μάλλον με την κυβέρνηση Κωσοπεδίου, κύριε Φέιθ, Πώς βλέπετε τα πράγματα, το διοικητικό δυναμικό της περιοχής σε τι κατάσταση βρίσκεται και πόσο χρόνο χρειάζεται το κοσυβοπαίδιο μέχρι να πετύχει πλήρη ε, ε, αυτάρκεια. Ευχαριστώ. Τέλος ο κύριος Γιούρι έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Πολλά υπόθηκαν για την πολιτική σταθεροποίηση του κοσυφοπεδίου. Ξέρουμε αυτό ότι είναι κάτι που εξαρτάται από τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας ε, στο Κωσυφοπαίδιο. Όμως εδράζεται και στη συνεργασία μεταξύ ε, των αρχών και της κοινωνίας των πολιτών. Επισκέφθηκα το Κωσυφοπαίδιο πριν ε, ανακηρυχθεί ανεξάρτητο και συμμετείχα σε μια διάσκεψη για την ε, ορθή πρακτική που ακολουθείται τη συμμετοχή των πολιτών στις, ε, δημόσιες, στα δημόσια πράγματα. Και ξέρω ότι έχουν πολύ ανεπτυγμένη κοινωνία των πολιτών. Έχουν πάνω από 3.000 καταχωρημένες μη κυβερνητικές οργανώσεις. Άρα υπάρχει ενδιαφέρον ε, για την οργανωμένη λειτουργία της κοινωνίας. Όμως παρατήρησα ότι υπάρχει και διαφορά μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών δηλαδή μεταξύ κοινωνίας των πολιτών και κοινοβουλίου και κοινωνίας πολιτών και κυβερνήσεως. Και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσο έχει επιτευχθεί κάποια πρόοδο στον τομέα, διότι εκφράστηκε η ευχή από τις μη κυβερνητικές οργανώσεις αυτή τη διάσκεψη. Ποια ευχή, ότι θα πρέπει να δημιουργηθούν κάποιοι μηχανισμοί που θα επιτρέπουν πιο άμεση συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στα τεκτενόμενα. Η κοινωνία των πολιτών είναι καλοργανωμένη, και δεν βασίζεται αποκλειστικά σε εθνοτικές βάσεις, υπάρχουν και μικτές μορφές συμμετοχίες Είναι πολύ καλές πρακτικές που ακολουθούνται που θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Ευχαριστώ. Κύριε Φέιθ, έχετε το λόγο. Για να απαντήσει σε αυτό το δεύτερο γύρο των συζητήσεων, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομο. Να επανέλθω στο θέμα των Ρωμά, που δεν αντιμετώπισα στην πρώτη στον πρώτο γύρο συζητήσεων. Τα μέτρα επίγουν. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Αυτό που με απογοητεύει κάπως είναι η σύγχυση ευθυνών των διαφόρων εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση της κατάστασης των Ρωμά. Όπως σας είπα, μας προβληματίζει η έλλειψη εύκολης πρόσβασης στον βορρά όπου βρίσκονται τα περισσότερα κέντρα φιλοξενίας των Ρωμά που έχουν διωχθεί. Να σας πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει την κατάσταση και έχουμε συμβάλει και υπάρχει σημαντική συμβολή και του ΠΟΗ και του USAID, τον είπα, που προσπαθούν να μετακινήσουν, να επαναφέρουν μάλλον την κοινότητα των Ρωμά και να βελτιώσουν την κατάστασή τους. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλουν να περάσουν την άλλη πλευρά του Ιμπαρ, το τον νότο, θέλουν να βρουν εναλλακτική λύση. Μπορώ να σας πω πάντως ότι είναι ένα σημαντικό θέμα που το προσέχουμε ιδιαίτερα. Um, uh, για τον κύριο Μέγερ, καταλαβαίνω τις uh, επιφυλάξεις που εκφράζεται για το κατά πόσο μπορούμε να έχουμε μια πολυεθνική κοινωνία. Πιστεύω ωστόσο ότι αυτή είναι, αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να προχωρήσουμε. Είχα την ευκαιρία να δουλέψω στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας Το παράδειγμα εφαρμόστηκε εκεί. Δεν υπάρχει δυνατότητα άλλη διατήρηση των χωρών αυτών με την εθνοτική σύνθεση που έχουν. Στόχος μας πρέπει να είναι να κρατήσουμε αυτή την πολυεθνικότητα και να προχωρήσουμε αργά-αργά ε, προς μια συμφιλίωση και βιώσιμη κατάσταση για όλες τις κοινότητες στην ε, χώρα. Η Μάλλον οι εναλλακτικέ λύσει θα ήταν η αστάθεια, θα ήταν ει βάρο της Ένωσης, θα ήταν αποτυχία και διάλυση των κρατών και επανάληψη της βίας. Το πιο σημαντικό ωστόσο είναι ότι μιλάμε για ευρωπαϊκές αξίες. Και στα κράτη-μέλη μας υπάρχουν μειονοτικές κοινότητες και τα μέλη, τα, τα, τα υποψήφια μέλη καταλαβαίνουν ότι πρέπει να αναζητήσουν πολυεθνικές λύσεις. Αυτή είναι η απόφαση μου στο δίλημα που αναφέρατε. Η σερβική κοινότητα θέλει να συνεχίσει να προσβλέπει προς το Βελιγράδι. Η αλβανική κοινότητα θέλει πλήρη ανεξαρτησία. Πλήρης ανεξαρτησία Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Βρισκόμαστε ακόμα στην ε, ελεγχόμενη ανεξαρτησία. Δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει αυτή η φάση. Ε, και απαντάω εδώ και στην ερώτηση του κ. Νασάουερ για τη διοικητική ικανότητα της κυβέρνησης να μπορέσει να συνεχίσει αφού επιτευχθεί η πλήρης ανεξαρτησία και βγούμε από αυτό που εσείς περιγράψετε ως προτεκτοράτο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι βασικές προϋποθέσεις για να περάσουμε από τη μία φάση στην πλήρη ανεξαρτησία είναι η ύπαρξη σταθερότητας σε όλο το κοσυφοπαίδιο και ένα, ένας ενιαίος νομικός χώρος να υπάρχουν καλές σχέσεις γυτνίασης μεταξύ κοσφοπεδίου και γειτόνων και το κοσφοπέδιο και οι γείτονές του να μπορέσουν να συνεχίσουν την πορεία τους με εμπιστοσύνη προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο όρος προτεκτοράτο λοιπόν είναι προβληματικός για μένα. Αν δώσετε σε μια χώρα την προοπτική ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως μέρος της Ένωσης θα μπει, όχι ως προτεκτοράτο. Αυτό το περιμένουν οι άνθρωποι εκεί. Γυναίκες. Συγκεκριμένα παραδείγματα για το θέμα αυτό των γυναικών. Είχα μια επαφή με την κοινωνία των πολιτών στο Κωσφοπέδιο πρόσφατα το εκτίμησαν ιδιαίτερα. Θέλανε να συνεχίσουν αυτές οι επαφές. Η κατάσταση τώρα όπως έχει είναι ότι έχει τεθεί μια ποσόστοση ενός τρίτου για τους υποψηφίους σε δημοτικές εκλογές να είναι γυναίκες. Σε ό,τι αφορά τη θέση της ε, EULEX αλλά και πάλι πρέπει να σας πω ότι δεν είμαι εγώ ο εκπρόσωπος της EULEX, είναι ο στρατηγός Καμπονέτ. Νομίζω ότι προσπαθεί να εξασφαλίσει μεγαλύτερη παρουσία γυναικών στην επιχείρηση της EULEX. Βέβαια αυτό είναι ένα σημείο που τα κάτι μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη γιατί τα κάτι μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν ο αναπληρωτής διευθυντής της αστυνομίας στο Κοσφοπέδιο στην Πριστίνα είναι γυναίκα. Έχουμε λοιπόν ενθαρρυντικά στοιχεία. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε εδρεωμένες παραδόσεις στην κοσοβάρικη κοινωνία, αλλά υπάρχουν και θετικά στοιχεία που δείχνουν ότι οι γυναίκες είναι έτοιμες να αναλάβουν τις ευθύνες τους και μπορώ να δώσω πολλά παραδείγματα γυναικών που ασκούν σημαντικά λειτουργήματα σε διάφορους τομείς του βίου στην στο Κοσφοπέδιο και σε διάφορες θέσεις στην κοινωνία. Το θέμα της διαφθοράς είναι ένα ζήτημα το οποίο θα είναι ένα κομβικό εγχείρημα για την EULEX. Εδώ περιμένω λοιπόν να υπάρξει πρόοδος σε σύντομο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να γίνουν ή να περατωθούν οι απαραίτητες έρευνες και ανακρίσεις. Είναι θέμα, η δίωξη λοιπόν θέμα της ULEX και των δικαστικών αρχών να έρθουν όλα αυτά τα άτομα ενώπιον της δικαιοσύνης χωρίς να ασκούνται διακρίσεις εναντί αυτών. Δεν θα πρέπει να ολιστήσουμε σε μια συνέχιση της συζήτησης για το πόσοι Σέρβοι και πόσοι Αλβανοί έρχονται ενώπιον της δικαιοσύνης. Η δικαιοσύνη είναι τυφλή Πρέπει να αντιμετωπιστούν λοιπόν όλα αυτά τα θέματα προτεραιότητος και το μόνο κριτήριο το οποίο θα πρέπει να πριτανεύει είναι η απόδοση δικαιοσύνης. Νομίζω ότι έχω περίπου εξαντλήσει τα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί. Κάπου θέσατε ένα ερώτημα από τον κύριο Νασάρε για το για το χρονικό ορίζοντα της εντολής της EULEX. Αυτό έχει καταρχήν αποφασιστεί από το Συμβούλιο να διαρκέσει δύο χρόνια εντολή της, αλλά είναι σαφές ότι ή απαραίτητον θα μπορούσε να παραταθεί η εντολή της. Επομένως τρέχει από το 2000, τον Ιούνιο του 2008 μέχρι τον Ιούνιο του 2010. Για να είμαι ρεαλιστής, αν πετύχει όλους τους στόχους της EULEX μέχρι το έτος 2010, αυτό θα είναι θαύμα. Επομένως, σίγουρα θα υπάρξει μια αίτηση παράτησης εντολής της Ιουλέξ. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε να μιλήσω στην Επιτροπή σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Φέιτ. Και εμεί χαιρόμαστε για την πλήρη κάλυψη όλων των θεμάτων του κόσμου πεδίου Νομίζω ότι υπήρξε μια μεγάλη σύγκληση μεταξύ των απόψεων του Κοινοβουλίου και των δικών σας απόψεων. Εκτιμούμε το έργο σας. Θα τα παρακολουθήσουμε τα θέματα αυτά και ελπίζω θα σας ξαναδούμε και κλείνω και τις συνεδρίαση επιπλέον.